Αγαπητοί συνάδελφοι, ήρθε η ώρα νομίζω να ξεκινήσουμε, γιατί ήδη έχουμε καθυστερήσει λίγα λεπτά. Θα ξεκινήσουμε με το πρώτο σημείο της ημερήσης διάταξης, δηλαδή την έγκρισή της. Η κυρία Καρντίνη, σε συμφωνία με τους κοιόδης συγκητές, ζήτησε να αναβληθεί η ψηφοφορία του σημείου 7 της ημερήσιας διάταξης, ε, το σημείο 15, μέχρι το Σεπτέμβριο, προκειμένου να οριστικοποιηθούν οι συμβαστικές τροπολογίες και να ολοκληρωθούν οι συζητήσεις με τις πολιτικές ομάδες. Με αυτή την αλλαγή λοιπόν, την αναβολή της ψηφοφορίας του σημείου 7 της κυρίας Γκαρτίνη για τις 15 Σεπτεμβρίου, μπορούμε να την εγκρίνουμε. Σημείο 2. Ανακοινώσει του Πρόεδρου. Έχουμε σήμερα διερμηνία σε 22 γλώσσες και μάλιστα ο φάκελος της σημερινής συνεδρίασης διατίθεται μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικής συνεδρίασης από το ίντερνετ. Έχουμε μοιράσει, στείλει και ηλεκτρονικά τις συστάσεις των συντονιστών. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις θα τις θα θεωρηθούν ως συγκεκριμένες. Και περνάμε τώρα στο σημείο 4 Έχουμε μαζί μας την Υπουργό Περιβάλλοντος του Λουξεμβούργου, την κυρία Καρόλ Ντίσεμπουργκ. Την ευχαριστώ θερμά που ήρθε για να μας παρουσιάσει τις προτεραιότητες ε, της Προεδρίας του Λουξεμβούργου για το επόμενο εξάμενο. Και ευχαριστώ την Υπουργό Ντίσεμπουργκ για την προθυμία της ε, να έρθει, γιατί είναι σημαντικό να έχουμε την ανταλλαγή απόψεων ήδη από την αρχή του εξαμήνου της Προεδρίας του Λουξεμβούργου. Θα σας δώσω το λόγο για μια εισαγωγική ομιλία και με, θα ακολουθήσει συζήτηση με τα μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτέ, κυρίες και κύριοι. Ειλικρινά αισθάνομαι περιχαρής για την ευκαιρία που έχουμε ε, να συζητήσουμε και να σας παρουσιάσω το πρόγραμμα και τις προτεραιότητες για το περιβάλλον ε, της ε, Προεδρίας του Λουξεμβούργου στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα θέματα που έχουμε στο μενού της Προεδρίας μας ε, εξαρτώνται φυσικά από τις νομοθετικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή αυτές που προτίμησε να αποσύρει. Προσωπικά οφείλω να ομολογήσω ότι απογοητεύτηκα εκτρά από το πρόγραμμα εργασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2015. Το νομοθετικό πακέτο για την κυκλική οικονομία, για παράδειγμα, αποσύρθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το πρόσχημα ότι ήταν αδύνατο να επιτευχθεί συμφωνία. Ενώ μόλις είχαν ξεκινήσει οι εργασίες ε, στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Για το θέμα αυτό θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη δική σας ε, στράτευση και δέσμευση, γιατί η κυκλική οικονομία δημιουργεί μια τεράστια ευκαιρία στην οικονομία μας ε, προκειμένου να καταστεί πιο ανταγωνιστική και να δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης. Η νέα πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναμένεται για το φθινόπωρο, προς το τέλος δηλαδή της Λουξεμβουργιανής Προεδρίας, θα μεριμνήσουμε ώστε να αναβαθμιστούν οι φιλοδοξίες της νέας πρότασης και να μην περιοριστούν μόνο σε μια διεύρυνση των αρμοδιοτήτων μεταξύ επιτρόπων. Και το επίπεδο περιβαλλοντικής φιλοδοξίας θα θέλαμε να ενισχυθεί. Μάλιστα, ε, έλαβα δεόντως υπόψη το σχετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που υιοθετήθηκε στις 9 Ιουλίου στην Ολομέλεια στο Στρασβούργο. Και θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια την κυρία Σύρπα Πιτεκάινεν και τους και εισηγητές ε, για την εξαιρετική εργασία τους. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει τις ίδιες προτεραιότητες και στόχους με την Προεδρία του Λουξεμβούργου για το θέμα αυτό. Τώρα επανέρχομαι στο νομοθετικό πακέτο. Η ποιότητα του αέρα και η σχετική οδηγία για τα εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών είναι από τις προτεραιότητες μας για το επόμενο εξάμεινο. Η πρόταση για τα εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών θα διαδραματίσετε με λιώδη ρόλο στην καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρήπανσης και στη μείωση των πρόωρων θανάτων που σχετίζονται με αυτή την ατμοσφαιρική ρήπαση. Και παρόλο που οι αντιπροσωπείες ε, ακόμη ε, εξετάζουν τις ε, προσωμιώσεις που έκανε η ΙΑΣΑ, δηλαδή το Διεθνές Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Ανάλυσης Θυμάτων, Πιστεύουμε ότι θα καταφέρουμε να απεμπλέξουμε την κατάσταση και να ξεπεράσουμε τα εμπόδια. Θα συνεχίσουμε λοιπόν την εξέταση αυτής της πρότασης και ε, την εξέταση των τροπολογιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου να διερευνήσουμε τις δυνατότητες σύναψης συμφωνίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μάλιστα στο εγγύς μέλλον. Η πρόταση του κανονισμού για τη μείωση των ρήπων των οδικών χυμάτων, δηλαδή το πρότυπα Euro 5 και 6, είναι ένα άλλο θέμα που εντάσσονται στο πλαίσιο της βελτίωσης της ποιότητας του αέρα. Έχω επίγνωση ότι η συμφωνία των εθνικών εταίρων γύρω από τις ε, εκπομπές σε συνθήκες ε, ε, πραγματικής ε, οδήγησης ε, θα μας ε, επιτρέψουν να ενισχύσουμε και να ολοκληρώσουμε τις προσπάθειές μας και δεν θα μας εμποδίσουν καμία περίπτωση. Ε, νομίζω ότι τέτοιες αποφάσεις θα πρέπει να ληφθούν από τους συνομοθέτες και όχι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό εξουσιοδότηση και χώρες εξουσιών, ιδιαίτερα για το καθορισμό των οριακών τιμών. Οπότε θα προσέξουμε ιδιαίτερως στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίως ε, την ψηφοφορία στην Επιτροπή Περιβάλλοντος ε, της 23 Σεπτεμβρίου. Και ανάλογα με το αποτέλεσμα και τις προθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά τη συνέχεια που θα δοθεί στο θέμα αυτό, η Προεδρία του Λουξεμβούργου είναι έτοιμη ε, να συνεργαστεί μαζί σας για να διερευνήσουμε τις δυνατότητες που υπάρχουν για τις περαιτέρω διαπραγματεύσεις. Είναι προφανές ότι τα θέματα για την ε, ποιότητα του αέρα είναι αλληλένδετα με τα ζητήματα του κλίματος, άλλη προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Προεδρίας και στο πλαίσιο αυτό η πρόταση για την ε, μεταρρύθμιση του συστήματος εμπορίας εκπομπών του ETS ε, γίνεται σήμερα ουσιαστικά. Ο Επίτροπος Αρίας Κανιέτε θα σας παρουσιάσει το απόγευμα την πρότασή του θα την παρουσιάσει και στο Συμβούλιο, στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος που θα λάβει χώρα στις 23 Ιουλίου. Θα ήθελα να χαιρετήσω και την ψηφοφορία που έγινε για το, για το αποθεματικό ε, αγοράς, ε, ε, για το αποθεματικό έκτακτο ανάγκης ε, και συγχαίρω τον Επίτροπο Κανιέτε που τήρησε την υπόσχεση του και το λόγο του. Η μεταρρύθμιση του συστήματος εμπορίας εκπομπών έχει θεμελιώδη σημασία και αποδεικνύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αναλαμβάνει δράση για να διασφαλίσει το ρόλο της, τον ηγετικό της ρόλο στην καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Από ότι η Ευρωπαϊκή Προεδρία θα ξεκινήσει στις αρχές Σεπτεμβρίου τις εργασίες στην αρμόδια ομάδα εργασίας για το περιβάλλον. Βέβαια, οι επόμενες προεδρίες θα πρέπει να καταλήξουν σε συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σε ό,τι αφορά τις ε, μη νομοθετικές προτάσεις, ε, το Συμβούλιο υιοθέτησε τις, ε, τα συμπεράσματα για τη στρατηγική 2020 και για το πρασίνισμα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου στις 28 Οκτωβρίου 2014. Ένα χειρό μήνυμα για τις περιβαλλοντικές πτυχές και την αηφορία της στρατηγικής. Εξακολουθεί να ισχύει το μήνυμα αυτό και προβλέπουμε ότι στο Συμβούλιο Περιβάλλοντος που θα λάβει χώρα στις 26 Οκτωβρίου 2015 θα διεξαχθεί συζήτηση για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και τις επιζήμιες επιδοτήσεις, harmful, harmful subsidies. Αυτά τα θέματα θα βρεθούν στο επίκεντρο της συζήτησης. Η Προεδρία του Λουξεμβούργου στο Συμβούλιο αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην προστασία και τη διαφύλαξη της βιοπικιλότητας στην Ευρώπη αλλά και παγκοσμίω και άρα στην εφαρμογή μιας αποτελεσματικής στρατηγικής. Και φυσικά παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς και τις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ιδιαίτερα τις συζητήσεις που γίνονται στα πλαίσια της έκθεσης πρωτοβουλίας του κυρίου Μέκερ και θα προτείνουμε το Δεκέμβριο στο Συμβούλιο την υιοθέτηση συμπερασμάτων που θα εμπνευστούν από την ενδιάμεση αναθεώρηση της ε, στρατηγικής για τη βιοπικιλότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, κάτι που έχει, ε, μας έχει υποσχεθεί το αργότερο για τα μέσα Οκτωβρίου ο Επίτροπος Βέλα. Σημαντική βάση αυτή για τις εργασίες, γιατί θα έχουμε και την υιοθέτηση της έκθεσης State of Nature της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος. Και με όλα αυτά τα συμπεράσματα θέλουμε να συμβάλλουμε στην υλοποίηση των έξι στόχων της στρατηγικής ε, για το 2020, διαμορφώνοντας ένα σαφέστερο πλαίσιο για την πρόοδο που έχει επιτελεστεί και κυρίως για αυτή που θα πρέπει να υλοποιηθεί στο μέλλον. Και περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον και την απαραίτητη απόσταση, τη, τα αποτελέσματα του εγχειρήματο REFIT ε, που γίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη συνέχεια που θα δοθεί στις οδηγίες για, το, για τα ενδιατήματα και τα πτηνά. Και ερχόμαστε τώρα στις ε, μείζονες προκλήσεις ε, παγκοσμίω και το πολυμερές ε, πρόγραμμα των Ηνωμένων Αθηνών για το 2015. Ε, μετά την διάσκεψη κορυφής για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης που γίνεται αυτή τη μέρε στην Αδισαμπέμπα, Έχουμε το Σεπτέμβριο στη Νέα Υόρκη την ειδική ε, σύνοδο Κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για την αηφόρο ανάπτυξη προκειμένου να καθοριστεί το πρόγραμμα για μετά το 2015 και τέλος έχουμε και την ε, διεθνή διάσκεψη κορυφή που θα γίνει στο Παρίσι, την COP21, για το περιβάλλον. Το πρόγραμμα τη αιφόρο ανάπτυξη για την περίοδο μετά το 2015 θα πρέπει να είναι αλληλέγγυο και να συνάδει με τους κλιματικούς στόχους. Η έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών ανταποκρίνεται στις προσδοκίες μας, ε, επανεπιβεβαιώνει το στόχο ε, των δύο βαθμών Κελσίου και την ημί υπέρβαση αυτού του στόχου και την ανάγκη ε, ανάπτυξης οικονομικής που θα προσαρμόζεται στις κλιματικές αλλαγές. Είναι σημαντική η περιβαλλοντική διάσταση για να ελοπίσουμε και το στόχο της εξάλληψης της φτώχειας, γιατί οι πλέον άποροι είναι αυτοί που πλήττονται περισσότερο από την ρήπανση και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα λοιπόν για μετά από το 2015 είναι προτεραιότητα του Ευρωπαϊκού της Προεδρίας του Λουξεμβούργου στο Συμβούλιο και το άτυπο Συμβούλιο Περιβάλλοντος 22 και 23 Ιουλίου θα αφιερωθεί στις συζητήσεις για τους περιβαλλοντικούς στόχους ε, με τον κύριο Άχιμ Στάινερ από το πρόγραμμα περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών. Όπω ξέρετε κύριε Πρόεδρε, βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη στιγμή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το περιβαλλοντικό κεκτημένο αυτή τη στιγμή διατρέχει κίνδυνο εξαιτία τη απορρίθμιση και τη τάση επανεθνικοποίηση. Θα πρέπει λοιπόν να, συνεργαστούμε στενά για να αποδείξουμε ότι οι πολιτικέ του περιβάλλοντο βελτιώνουν το βιωτικό επίπεδο και την ποιότητα ζωή των Ευρωπαίων πολιτών και ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία της οικονομίας μας. Στην καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών θα πρέπει να είμαστε υπερήφανοι για τα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να γίνουμε υπόδειγμα για τους άλλους. Και ερχόμαστε στο κύριο θέμα της Προεδρίας μας, την 21η Σύνοδο της Διάσκεψης των Μερών της ε, Σύμβασης Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις Κλιματικές Αλλαγές, COP21. Στις ε, 28 Σεπτεμβρίου το Συμβούλιο θα υιοθετήσει τα συμπεράσματα εν ώψη της προετοιμασίας της COP21 και θα προσπαθήσουμε να διαμορφώσουμε την πιο φιλόδοξη εντολή εν ώψη της COP21, γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ότι θα πρέπει να καταλήξουμε στο Παρίσι σε μια φιλόδοξη συμφωνία, ώστε να υιοθετήσουμε σωρό το όριο την αύξηση κατά δύο βαθμούς Κελσίου. Από την άποψη αυτή η συμφωνία θα πρέπει να καθορίζεται από ένα μακροπρόθεσμο όραμα της μετάβασης σε μια κοινωνία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια νομικά δεσμευτική συμφωνία, βιώσιμη και δυναμική, για να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων, ε, μια συμφωνία που θα αφορά το μετριασμό των κλιματικών συνθήκων και τον τρόπο ε, εφαρμογή των πολιτικών για να υλοποιήσουμε το στόχο. Θέλουμε ξεκάθαρου κανόνε και μια διαδικασία εφαρμογή του. Μόνο μια τέτοια συμφωνία όλων των μερών δεσμευτική θα δώσουμε ένα χειρό μήνυμα προ όλου του ε, παράγοντε και φορεί, όχι μόνο του κυβερνητικού, αλλά και τι επιχειρήσει, μη κυβερνητικέ οργανώσει και την τοπική αυτοδιοίκηση. Η πρόσφατη δήλωση του G7 τον Ιούνιο ήταν ένα πολύ ενθαρρυντικό μήνυμα ότι το μήνυμα ε, έγινε δεκτό στο υψηλότερο επίπεδο ή έφτασε μάλλον στο υψηλότερο επίπεδο. Γι' αυτό και η Προεδρία του Λουξεμβούργου θα επικεντρωθεί στις κλιματικές αλλαγές που είναι σημείο κλειδί για να καταλήξουμε σε καλή συμφωνία στο Παρίσι. Γι' αυτό και το θέμα του περιβάλλοντος θα αποτελέσει προτεραιότητα και θα συζητηθεί και σε υπουργικό επίπεδο ε, και στα Συμβούλια Περιβάλλοντος και στα Συμβούλια Υπουργών Οικονομικών. Επίσης, είμαστε υπέρ της ιδέας μιας εργαλειοθήκης με ένα ευρύ πρόγραμμα χρηματοπιστωτικών ε, μέσων δημόσιο και ιδιωτικού τομέα. Και πριν περάσουμε στη συζήτηση για να ακούσω τις ερωτήσεις σας, θα ήθελα να σας επισημάνω ότι κάποια από τα θέματα που σας απασχολούν δεν εμπίπτουν στο δικό μου χαρταφυλάκιο για παράδειγμα τα θέματα υγείας των ανθρώπων, υγείας των ζώων, ασφάλειας των τροφίμων. Αυτά τα θέματα θα σας τα παρουσιάσει αύριο ο υπουργό Υγείας. Εγώ θα βάλω τα δυνατά μου για να προωθήσω τα θέματα αρμοδιοτήτων μου και ήδη χαίρομαι εκ των προτέρων για τη συνεργασία που θα έχουμε με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τους επόμενους μήνες και σας ευχαριστώ θέρμα για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την εισήγησή σας και τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε με τον πρώτο γύρο ερωτήσεων με τους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων ο Ιβο Μπέλετ από το ΕΛΚ. Σας ευχαριστώ Κυρία Υπουργέ, θα σας κάνω κάποιες ερωτήσεις. Καταρχήν, διαπιστώνουμε ότι η φιλοδοξία σας για την κυκλική οικονομία είναι αρκετά ψηλή. Σας στηρίζουμε 100%. Και στο Κοινοβούλιο και σίγουρα σε αυτήν εδώ την Επιτροπή δεν μπορείτε να βασιστείτε στην βοήθειά μας και την πίστη μας για να πιέσουμε την Κομισιόν ώστε να προχωρήσει σε ένα φιλόδοξο, με αυτό μάλλον το φιλόδοξο πρόγραμμα. Είπατε ότι είναι το κύριο πιάτο η διάσκεψη για το κλίμα στο Παρίσι, υπό τη δική σας Προεδρία. Και ελπίζουμε ότι όλα αυτά θα ολοκληρωθούν με επιτυχία. Δεν ξέρω αν είναι τύχη, αλλά είπατε σήμερα ότι, το είπατε κι εσείς μάλλον, σήμερα ο, ο Επίτροπος Κανιέτε θα υποβάλει πρόταση για την αναθεώρηση του συστήματος ETS ε, διότι ο τομέας της ε, βιομηχανίας και της ενέργειας θα πρέπει να συμβάλλει σημαντικά μέχρι το 2030, ώστε να εγγυηθούμε μια μείωση της τάξης του, 40% ε, του διοξιδίου του άνθρακα. Κάποιες ερωτήσεις σχετικά. Τι γνώμη έχετε για τις προσπάθειες του τομέα της ε, αεροπλοείας και της ναυσιπλοείας, γιατί έχουν ακόμα δρόμο μπροστά τους αυτοί οι δύο τομείς. Προσπαθούμε να συνάψουμε μια διεθνή συμφωνία πριν το τέλος του επόμενου έτους και αυτό περιλαμβάνεται και στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου. Κατά τη γνώμη σας, αν ε, αυτό δεν λειτουργήσει σε διεθνές επίπεδο, ποιες θα είναι οι συμφωνίες που θα πρέπει να ε, συναυθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το τομέα της ναυσιπλοείας και της αεροπλογίας. Για το ETS και το μη, ε, και, και το μη ETS, ποιος θα πρέπει να καταβάλει τις πιο σημαντικές προσπάθειες και ποιος θα μπορούσε να κάνει ακόμα περισσότερο, γιατί το ETS, η ενέργεια και η βιομηχανία θα πρέπει να κάνουν ένα κομμάτι της προσπάθειας, αλλά υπάρχει και η διεθνής ε, διάσκεψη που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη και τα συμφέροντα της βιομηχανίας μας που δεν πρέπει να την διώξουμε από την Ευρώπη. Ε, να σκεφτούμε ακόμα την διαρροή άνθρακα, carbon leakage. άλλοι τομείς θα μπορούσαν να κάνουν πιο σημαντική προσπάθεια. Και η αντιστάθμιση σε σχέση με τις αναπτυσσόμενες χώρες, το offset, θα ήταν ίσως μια ενδιαφέρουσα ιδέα για να μπορέσουμε να τροφοδοτήσουμε το κλιματικό ταμείο. Τέλος, ε, ε, Κύριε Υπουργέ, αναφέρατε την οδηγία Habitat και τη διάδοχό της, ε, την βιοπικιλότητα που απειλείται σε πολλά μέρη της Ένωσης. Ποια είναι η δική σας ε, εικόνα, η οδηγία Habitat θα πρέπει να μείνει ως έχει, αλλά να εφαρμοστεί καλύτερα ή μήπως θα έπρεπε να τολμήσουμε να ζητήσουμε από την Κομισιόν να αναθεωρήσει την οδηγία Habitat και να υποβάλει πρόταση τροποποίησης της οδηγίας αυτής καθώς ε, υπάρχει εντύπωση ότι για κάποια είδη χρειάζεται καλύτερη προστασία. Αλλά είναι δύσκολο να συνεργαστούμε σε κάποιες ε, περιοχές με τη γεωργία και με την βιομηχανία. Εσείς ε, τι εικόνα έχετε για αυτή την ισορροπία και πώς θα μπορούσαμε να ε, αναθεωρήσουμε την οδηγία αυτή. Σοσιαλιστές Ματίας Γκρότ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Υπουργέ, προσβλέπω στην Προεδρία του Λουξεμβούργου, διότι όλα αυτά που λέτε μας υπόσχονται πολλά. Συζητήσαμε με την ε, Επίτροπο το θέμα του Ρίφιτ, ε, με την... συζητήσαμε την προστασία της ε, φύσης των βιότοπων στην Ευρώπη. Δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα και κατά τη γνώμη μου θα ήταν τελείως ε, λάθος ε, νόημα αν ε, ξανανοίγαμε όλο το πακέτο αυτό. Η γερμανική κυβέρνηση έχει διαφωνήσει με το άνοιγμα του θέματος αυτού. Έχετε την δυνατότητα να εκτόσετε συμπεράσματα του Συμβουλίου και θα δούμε προς ποια κατεύθυνση θα πάνε τα πράγματα. Ε, κατόπιν έχουμε την οδηγία για τον ε, καθαρό αέρα. Οι ε, πρόοροι θάνατοι που είχαμε νομίζω ότι αρκούν το θέμα αυτό είναι δική σας αρμοδιότητα. Όσον αφορά την αμμονία και το μεθάνιο θα πρέπει να συζητήσουμε τα θέματα αυτά περαιτέρω και να ασκήσουμε δημοσίως πίεση. Χρειαζόμαστε καλή νομοθεσία στον τομέα αυτών. Θα με ενδιέφερε λοιπόν να γνωρίζω πόσο έχει προχωρήσει η συζήτηση στο Συμβούλιο. Υπήρξαν δυσκολίες, μπορούμε να τις ξεπεράσουμε. Οι 4.000 πρόοροι θάνατοι θα πρέπει να μειωθούν, διότι κατά τη γνώμη μου είναι σκάνδαλο σε μια κοινωνία κρατών όπως είναι η Ευρώπη να μην είναι δυνατόν να μειωθεί αυτός ο αριθμός. Αντιθέτως, τα τελευταία χρόνια ε, συνεχώς αυξάνεται αυτά πολύ σύντομα. Στην διάσκεψη COP θα συζητήσουμε το κλίμα. Και για το Κοινοβούλιο θα είναι κεντρικό θέμα αυτό που θα παρουσιαστεί σήμερα το απόγευμα, το σύστημα εμπορίας εκπομπών. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πόσο θα προχωρήσει το Κοινοβούλιο στο θέμα αυτό, εάν θα υποβάλει φιλόδοξη πρόταση, διότι αλλιώς βλέπω τον κίνδυνο στο μέλλον να έχουμε πρότυπα για εργοστάσια παραγωγής ενέργειας ε, τα οποία να μην ε, αρκούν. Επίσης όσον αφορά τον άνθρακα, και τον ψευδάργυρο βλέπουμε σε μελέτες πόσος ε, ε, υδράργυρο συγγνώμη, εκπέμπεται από ε, την παραγωγή ενέργειας από άνθρακα στην Ευρώπη. Είναι σκανδαλώδες αυτό, θα πρέπει λοιπόν να το ρυθμίσουμε. και αν δεν αρκούν τα μέτρα που θα ληφθούν ε, θα πρέπει να προχωρήσουμε σε περαιτέρω νομοθετήματα. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Κέρινγκ από το ECR. Α, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Υπουργέ, θα ήθελα εκ μέρους ε, της ομάδας ε, του ECR να σας ε, καλωσορίσω στην Επιτροπή μας. Αναφερθήκατε στην έκθεση πρωτοβουλίας για την ενδιάμεση αναθεώρηση της στρατηγικής βιοπικιλότητας. Είμαι εισηγητής για το θέμα αυτό και γι' αυτό θα ήθελα να μιλήσω για το θέμα αυτό και να σας θέσω κάποιες ερωτήσεις. Επιλέξατε πολύ καλό σύνθημα για την Προεδρία σας, Ένωση Πολιτών. Χαίρομαι λοιπόν που το Λουξεμβούργο, η Προεδρία του Λουξεμβούργου τονίζει ακριβώς το ρόλο των πολιτών. Εάν κάτι χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή, τώρα που η πίστη του κοινού βρίσκεται κάτω από το μηδέν, θα πρέπει να δείξουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση λαμβάνει υπόψη τους πολίτες και την θέση τους το πρόβλημα της βιοπικιλότητας και της προστασίας της φύσης είναι κάτι που ενδιαφέρει τους πολίτες μας. Είναι κάτι που τους, κάνει να... τους ανησυχεί τόσο πολύ που ξαγρυπνούν για το θέμα αυτό. Είχαμε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο λειτουργεί πολύ καλά. Ο κόσμος δεν θέλει να δει να αποδυναμώνεται η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτών. Η πρώτη μου ερώτηση λοιπόν είναι το μήνυμα αυτό των εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών πώς μπορείτε να διασφαλίσετε ότι θα ληφθεί υπόψη. Επίσης, Είμαι περίεργος να μάθω ποιο είναι το όραμά σας για τον τομέα αυτόν. Εάν εφαρμοστεί σωστά η ευρωπαϊκή νομοθεσία, μερικές φορές βλέπουμε θεαματικά αποτελέσματα. Το αποτέλεσμα εδώ θα είναι μεγάλη αύξηση της βιοπικιλότητας. Σε κάποια κράτη-μέλη όμως η εφαρμογή είναι ελλειπής. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω ποια είναι η θέση σας για το θέμα αυτό. Ε, σηκώσατε λίγο την άκρη του πέπλου πριν, διότι αναφερθήκατε στην ενδιάμεση αναθεώρηση για το στρατηγικό σχέδιο βιοπικιλότητας. Εγώ θα ήθελα να έχω περισσότερα στοιχεία. και να μάθω ποιες είναι οι φιλοδοξίες της Προεδρίας σας στον τομέα αυτών. Ελπίζω ότι θα συνεργαστούμε στενά μαζί σας και σας εύχομαι κάθε επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Ε, η ο κύριος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, ευχαριστώ κυρία Υπουργέ για την πολύ φιλόδοξη εισήγησή σας. Νομίζω ότι στον τομέα μας η δυσκολία είναι ότι οι πιο σημαντικές αποφάσεις στον τομέα μας δεν λαμβάνονται από εμάς ή τους υπουργούς ε, περιβάλλοντος, αλλά από άλλους ευρωβουλευτές και άλλους υπουργούς. Αυτό το γνωρίζετε πολύ καλά. Επικροτώ λοιπόν το γεγονός ότι οργανώνεται αυτό το κοινό συμβούλιο για την ε, οικονομική πλευρά της περιβαλλοντικής πολιτικής και προσβλέπω στα αποτελέσματα αυτού του συμβουλίου. Ε, το πρόβλημα όμως δεν βρίσκεται μόνο στον τομέα του κλίματος, ε, βρίσκεται και σε άλλους τομείς. Θα επικεντρωθώ λοιπόν ακριβώς σε αυτό. Αν εξετάσουμε την κυκλική οικονομία και τη συζήτηση που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα στο Κοινοβούλιο, ο Επίτροπος Βέλα δεν ήταν παρόν στο ημικύκλιο. Είχαμε τους δύο αντιπροέδρους, Τίμερμανς και Κατάινεν, που είναι αρμόδιοι για την οικονομική πολιτική μας. Πιστεύω ότι αυτό είναι πολύ θετικό μήνυμα. Η έκθεση McKinsey που παρουσιάστηκε στις ε, 25 Ιουνίου αναφέρεται ε, στα κέρδη από την κυκλική οικονομία, τα οποία ανέρχονται σε εκατομμύρια, όχι μόνο δισεκατομμύρια. Θεωρούν ότι η κυκλική οικονομία θα πρέπει να είναι το επόμενο σημαντικό ευρωπαϊκό οικονομικό εγχείρημα. Είσαστε λοιπόν διατεθμένοι να οργανώσετε μαζί με το Συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ μία συνάντηση για την κυκλική οικονομία, διότι νομίζω ότι τα περιβαλλοντικά ωφέλη αποτελούν πολύ ωραία παρενέργεια ε, της κυκλικής οικονομίας, την οποία όμως χρειαζόμαστε για οικονομικούς λόγους. Και τέλος, ε, κύριε Πρόεδρε, η τελική μου παρατήρηση έχει να κάνει με την ε, βιοπικιλότητα. Είδαμε την έκθεση State of Nature και το βασικό συμπέρασμα είναι ότι δεν κάνουμε αρκετά ακόμα. Διαφωνώ λοιπόν ριζικά με την ερώτηση του Ιβου Πελέτ. Δεν θα πρέπει να αποδυναμώσουμε, δεν θα πρέπει να ξανανοίξουμε το θέμα των ε, ε, οδηγιών μας για τους βιότοπους και για τα πτηνά. Θα πρέπει να σκεφτούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε την κατάσταση της φύσης σε σχέση με τώρα. Και ένα από τα προβλήματα που επεσήμανε η έκθεση State of Nature ήταν η γεωργία. Η εντατική γεωργία θεωρείται ε, μία από τις βασικές αιτίες για την απώλεια βιοπικιλότητας. Ξέρουμε ότι η κοινή γεωργική πολιτική δεν αποτελεί μεγάλη επιτυχία. Η αρχική πρόταση της Κομισιόν αποδυναμώθηκε σε μεγάλο βαθμό από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι, είστε διατεθειμένοι να αγωνιστείτε για αναθεώρηση της κοινή γεωργικής πολιτικής έχοντας υπόψη την, ε, έχοντας κατά νου την βιοπικιλότητα και τέλος ε, κύριε Πρόεδρε, η κυρία Υπουργός συμφωνεί μαζί μου ότι οι γεωργικές αποφάσεις λαμβάνονται σε κενό αέρος και όχι από την Κορεπέρ. Δηλαδή έχουμε εδώ έναν απομονωμένο τομέα όπου λαμβάνονται αποφάσεις και νομίζω ότι αυτό είναι ένας λόγος που οι αποφάσεις που λαμβάνονται εκεί δεν ωφελούν το σύνολο της κοινωνίας. Ευχαριστώ. Ε, Také mě dovolte paní ministrní hodně úspěchu, protože priority, které nám i tady dnes... Ευχαριστώ. Και εγώ θέλω να σας ευχηθώ καλή επιτυχία γιατί οι προτεραιότητες που μας ε, εκθέσατε σήμερα είναι εξαιρετικά φιλόδοξες. Και για μας επίσης είναι πολύ σημαντικό ε, να οργανώνονται τέτοιου είδους πράγματα γιατί μας μένουν τέσσερις μήνες για το ETS. Και πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό γιατί ε, στο τέλος θα έχουμε τη διάσκεψη του Παρισιού που, για την οποία ευχόμαστε καλή επιτυχία επίσης και όπου και ελπίζουμε ότι τα μισή τουλάχιστον αυτών των προτεραιοτήτων θα έχουν υλοποιηθεί μέχρι το Δεκέμβριο. Τι γίνεται με τα ανώτατα εθνικά όρια, γιατί η ψηφοφορία στο Ευρωκοινοβούλιο θα γίνει τέλη Οκτωβρίου. Θα ήθελα να γνωρίζω λοιπόν ποιο είναι το επόμενο στάδιο. Με το τρίλογο και τα λοιπά. Τι προετοιμάζει το Συμβούλιο και ποια θα είναι η θέση σας στο πλαίσιο αυτών των εθνικών ανώτατων οριών για τις εκπομπές ψηφία του άνθρακα. Ένα άλλο θέμα το οποίο είναι τμήμα των αρμοδιοτήτων μας, είναι η ενημέρωση και η προστασία των καταναλωτών, ένα σημαντικό θέμα αυτό, γιατί στις μελέτες διαπιστώνουμε ότι οι καταναλωτές συχνά απογοητεύονται ε, ε, ή ακόμα και βλάπτεται η υγεία τους. Θα πρέπει ίσως να εστιαστούμε σε αυτό το θέμα στη διάρκεια της Προεδρίας σας. Ένα ακόμα θέμα το οποίο δεν έχουμε ακόμα αναφέρει. Γράφετε στο έγγραφο της Προεδρίας σας ότι θα προσπαθήσετε να συμβάλλετε στη δημοκρατική συζήτηση και στην αναθεώρηση των διατάξεων όσον αφορά τους μη τροποποιημένους οργανισμούς, γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Ε, Θα ήθελα να ξέρω αν, θα ανοίξετε αυτή τη συζήτηση εκ νέου. Θα ήθελα να γνωρίζω τη γνώμη σας. Και επίσης μιλήσατε για την συνεργασία που είναι απαραίτητη εν ώψη της ΚΟΠ στο Παρίσι. Αυτή τη στιγμή επικρατεί κάποιο ε, κάποια σύγχυση. Δεν ξέρουμε πώς θα διαπραγματευτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιος θα ηγηθεί, πώς θα είναι η συνεργασία ανάμεσα στους κεντρικούς φορείς που θα αποφασίσουν στο Παρίσι. Νομίζω πως αυτό είναι κομμάτι των αρμοδιοτήτων σας. Πώς θα οργανωθούν όμως όλα αυτά ανάμεσα στους θεσμούς πώς θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτούς τους φιλόδοξους στόχους στην πράξη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Από τους πράσινους. Ο κύριος Έκχαουτ. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ για την εισήγηση που μας κάνατε. Έχετε πολλά θέματα στην ατζέντα σας. Ενδιαφέρονται ήταν αυτοί οι έξι μήνες με τις διαπραγματεύσεις για την ποιότητα του αέρα, μάλλον την βιοπικιλότητα, ε, και την κυκλική οικονομία. Πολύ κρίσιμα και σημαντικά όλα αυτά τα θέματα. Προσβλέπω πραγματικά στη συνεργασία με την Προεδρία σας σε αυτά τα θέματα. Ένα από τα πιο σημαντικά όμως είναι φυσικά το Παρίσι στο τέλος του έτους και σε αυτό θέλω να εστιάσω τις ερωτήσεις μου. Αν δούμε την κατάσταση που βρίσκεται η Ένωση, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Ένωση προσφέρει κάτι αλλά σίγουρα θα αμφισβητηθούμε στο Παρίσι. Και θα ήθελα να γνωρίσω τη στρατηγική σας, πώς πιστεύετε ότι η Ένωση ε, στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων προς το Παρίσι αλλά και στο Παρίσι προετοιμάζεται για το more for more, περισσότερα για περισσότερα όταν αυτό χρειαστεί στη διαπραγματεύση. Γιατί ξέρετε πώς πάνε οι διαπραγματεύσεις. Ε, γίνεται μια προσφορά, μετά οι άλλοι ζητάνε και προσδοκούν κάτι από εμά και πάει λέγοντα το λάθος στην Κοπεχάγη ήταν ότι η Ευρώπη δεν ήταν έτοιμη για ευελιξία στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω πώ θα το κάνετε όλο αυτό. και πώς θα έχουν οι, τα πορίσματα. Αυτή, τη στιγμή με βάση τα πορίσματα του δεν μπορούμε να κινηθούμε στο Παρίσι. Χρειάζονται ακόμα κατά τη γνώμη μου τρία πράγματα και θέλω τη γνώμη σας. Καταρχήν την υπόσχεση μείον 20% το 2020, ενώ ξέρουμε ότι το έχουμε ήδη ξεπεράσει αυτό το στόχο σαν Ένωση. Πολύ εύκολο λοιπόν να προσφέρουμε περισσότερα πριν το 2020. Γιατί ήδη το έχουμε ξεπεράσει αυτό το στόχο. Προτίθεστε να ανοίξετε αυτή τη συζήτηση και στο Συμβούλιο Περιβάλλοντος. Δεύτερον, ε, χρειαζόμαστε μάλλον πενταετή ε, ε, αναθεώρηση. Ξέρω πως η Ένωση πάντοτε σκέφτεται το 30, αλλά οι διαπραγματεύσεις μιλάνε για πενταετής στόχους, ίσως λοιπόν και για πενταετή αναθεώρηση. Και επίση αυτό που είναι πολύ σημαντικό όταν συζητάμε στόχο του 2050 και η Ένωση που προσφέρει το μείον 60%, ξέρουμε πω αυτό το σενάριο συμφωνεί μόνο με του δύο βαθμού. Αν υπάρχουν τεράστιε αρνητικέ εκπομπέ αμέσω μετά το 2050. Και μιλάμε για τεράστιε αρνητικέ εκπομπέ. Μέχρι τώρα η Ένωση δεν είναι καθόλου προετοιμασμένη για το πώς θα επιτύχει αυτές τις αρνητικές εκπομπές. Πώς θα ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση, γιατί αν δεν έχουμε αυτές τις αρνητικές εκπομπές, η υπόσχεση της Ένωσης δεν συμφωνεί με τους δύο βαθμούς και αυτό δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Πάντως, όπως σας είπα, προσβλέπω σε μια ε, ξέρετη συνεργασία. Ευχαριστώ τώρα εξ ονόματος του FTD, ο κύριος Αφρόντε. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Τα δύο πιο σημαντικά σημεία για τους επόμενους μήνες, κατά τη γνώμη μου, είναι η COP21 και η οδηγία Habitat και πτηνά. Τα ανέφεραν όμως πολλοί συνάδελφοι και τα είπατε και εσείς στην εισήγησή σας, την οποία βρήκα πολύ ε, σαφή και σχετικά πλήρη σε σχέση με το χρόνο που έχετε στη διάθεσή σας για τη σχέση, στην έκθεση μάλλον για την ε, κατάσταση της φύσης. Ξέρουμε ότι αυτό βασίζεται ε, τα πορίσματα στα στοιχεία που έχουν ε, συγκεντρωθεί τα τελευταία χρόνια. Πάντως υπάρχει διαφορά ανάμεσα στα στοιχεία που έχουμε για, τα χερσαία, ε, για την κατάσταση της γης και σε σχέση με αυτά που έχουμε για τα, θάλασσα. Ε, τα στοιχεία για τη θάλασσα είναι λιγοστά και πρέπει να καταβληθούν πολλές περισσότερες προσπάθειες. Ε, το 60% είναι αρνητικό, αρνητικά τα στοιχεία που ξέρουμε και για τη Μαύρη Θάλασσα και για τη Βαλτική Θάλασσα, για να μην μιλήσουμε για την Μεσόγειο. Είδαμε την τελευταία έκθεση που η Κομισιόν ε, ανησυχεί ιδιαίτερα, εκφράζει ιδιαίτερε ανησυχίε για την Μεσόγειο. Στη Μεσόγειο και στη Μαύρη Θάλασσα τα ε, ε, στόκα αλευμάτων έχουν υπεραλλιευθεί και έχουν αλλιευθεί μάλιστα πέρα από το επίπεδο της βιωσιμότητας. Εγώ είμαι μέλος και της Επιτροπής Αλίας και είδαμε πόσο δύσκολο είναι να προσπαθήσουμε να επιβάλλουμε μια βιώσιμη αλληλεία ή τις περιβαλλοντικές οδηγίες χωρίς να έχουμε μια στέρεη ε, επιστημονική βάση με στοιχεία πλήρη ε, τα οποία να είναι επιστημονικώς ε, έγκυρα. Ακριβώς για τη θάλασσα αυτά τα στοιχεία λείπουν. Χρειάζονται πολύ σημαντικέ προσπάθειες έρευνας και συντονισμού για να μπορέσουμε να φτιάξουμε μια στέρεη βάση επιστημονικών στοιχείων για να μπορέσουμε εκεί να βασίσουμε τις πολιτικές μας και να βελτιώσουμε την κατάσταση των θαλασσών. Γι' αυτό σας ρωτώ. Τι θα κάνετε για να συμπληρώσετε αυτά τα κενά που έχουν συνέπειες σε όλες τις πολιτικές αποφάσεις που λαμβάνουμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Γιάλκα ε, από την ομάδα ΕΝΕΦ. Κύριε Υπουργέ, καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας. Δεν είναι καθόλου εύκολο το έργο σας, κύριε Υπουργέ. Γιατί κάθε φορά που μια νέα χώρα αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή κάθε εξάμεινο, οι αρμόδιοι υπουργοί έρχονται στις κοινοβουλευτικές επιτροπές και παρουσιάζουν τις προτεραιότητες της Προεδρίας τους. Ελπίζω λέγοντας ότι γενικώ κάθε εξάμεινο ακούμε τετριμένα και κοινοτοπίες ε, και ελπίζω να μην προσβάλλω τους προκατόχους σας. Ε, μας μιλάνε για ανταγωνιστικότητα, πρόθεση του οικολογικού χαρακτήρα, μεταρρυθμίση του συστήματος εμπορίας εκπομπών, ποιότητα του αέρα, ε, πρόοδος που πρέπει να γίνει στα μεταλλαγμένα, υποχρέωση να καταλήξουμε συμφωνία για τα ανατρόφιμα και τέλος ε, για τη συνδιάσκεψη των Παρισίων, COP21, που θα γίνει το Δεκέμβριο. Ε, τα βρίσκουμε όλα αυτά τα θέματα παντού και στις προτεραιότητες του Προεδρείου για το δεύτερο εξάμεινο του 2015. Στη Γαλλία όταν έχουμε τέτοια βουλημία φιλόδοξους στόχους λέμε όποιος, ε, όπου ακούς πολλά κεράσια κράτα και μικρό καλάθι. Ε, το θέμα είναι ότι ε, περισσότερο έχετε επικοινωνιακές φιλοδοξίες παρά αποφασιστικότητα και ελπίζω ε, να αφήσετε το στίγμα σας και να μην μείνετε σε απλά λόγια. Φυσικά θα πρέπει να εντάξουμε τις προτεραιότητες σε ένα πιο μακροπρόθεσμο σχέδιο για να αποφύγουμε τις συνέπειες ε, των διαδοχικών προεδριών. Ε, ακριβώς εξαιτία αυτή τη ε, πληθώρα των στόχων η αποτελεσματικότητα είναι περιορισμένη. Καλύτερα να περιοριστείτε σε μία, δύο, το πολύ τρει προτεραιότητε, Γιατί όλοι οι μεγάλοι στρατηγοί γνωρίζουν ότι για να κερδιθεί μια αποφασιστική μάχη θα πρέπει να επικεντρωθούν οι δυνάμει σε συγκεκριμένα σημεία. Και αυτή η στρατηγική θα μας επιτρέψει ε, να ξεκινήσουμε μια δυναμική που θα μας οδηγήσει στη νίκη. Ε, γιατί να μην τολμήσετε ε, να είστε πρωτότυποι, να επικεντρωθείτε σε λίγες προτεραιότητες και να αφήσετε τη, την πολυμορφία και την πληθώρα. Γιατί στην ε, Γαλλία 100 δισεκατομμύρια ευρώ είναι το κόστος της ατμοσφαιρικής ρήπανσης για να μην μιλήσουμε για την απώλεια της βιοπικιλότητας για το πλήγμα στην ανθρώπινη υγεία και στη γεωργία νομίζω πρέπει να επικεντρωθούμε στις ε, πιο φλέγουσες ανησυχίες των συμπολιτών μας αυτή τη στιγμή αντί να χανόμαστε σε πολλούς στόχους Μάλιστα Έγινε ένας πρώτος γύρος με εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων θα δώσω τώρα το λόγο στην εκπρόσωπο της Προεδρίας του Λουξεμβούργου, στην Υπουργό Ντίσπουργκ, για να μας δώσει απαντήσεις ε, στα θέματα που έθιξαν οι συνάδελφοι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ διότι τα περισσότερα από όσα άκουσα ήταν υποστήριξη για τις προσπάθειές μας. Ε, καταρχάς λοιπόν κύριε Μπέλετ, ναι, όλοι οι τομείς, η θάλασσα, ο, ο ναυτιλιακός τομέας δηλαδή, ε, η βιομηχανία θα πρέπει να συμβάλλουν. Θέσατε κάποιες ερωτήσεις, συμμεριζόμαστε τις ανησυχίες σας ε, και θα αναλύσουμε την ε, έκθεση το στομότερο δυνατών. Όπως και άλλοι αναφερθήκατε στην, ε, στις οδηγίες ευθυνών και βιοτόπων. Αυτοί είναι οι βασικοί πυλώνες της στρατηγικής μας για την προστασία της φύσης. Πιο σημαντικό είναι να εφαρμοστούν σωστά, διότι μας ε, παρέχουν ε, κάποια ασφάλεια σε νομικό επίπεδο. Και θα επαναλάβω αυτό που ήδη είπε ο Ματίας Γκρότε. Είπατε ότι όπου εφαρμόζεται σωστά η νομοθεσία βλέπουμε καλά αποτελέσματα. Πιστεύουμε λοιπόν ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε στην σωστή εφαρμογή και να μιλήσουμε και για τις πολιτικές χρηματοδότησης. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τις δικές σας ερωτήσεις. Προχωρώ στις ερωτήσεις του Ματίας Γκρότε. Αναφερθήκατε στην βιοπικιλότητα. Χαίρομαι για την επιστολή που εστάλει και θα προσπαθήσουμε στα συμπεράσματά μας να διαπιστώσουμε τι έχουμε αυτή τη στιγμή. Διαπιστώνουμε ότι όπου εφαρμόστηκαν σωστά οι οδηγίες έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα. Νομίζω λοιπόν ότι συμφωνούμε στο θέμα αυτό. Το δεύτερο θέμα στο οποίο αναφερθήκατε ήταν ε, ο αέρας, η ποιότητα του αέρα. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να προωθήσουμε την σχετική οδηγία. Η τελευταία συζήτηση που είχαμε στο Συμβούλιο ήταν ακριβώς ένα περαιτέρω βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Είχαμε επίσης κάποιες ερωτήσεις για την ε, βιοπικιλότητα. Ήδη αναφέρθηκα για τη θέση της Προεδρίας. Είναι σαφής η θέση της Προεδρίας. Σας ευχαριστώ για την παρατήρησή σας και προσβλέπουμε στην καλή συνεργασία μαζί σας. Και ναι, πράγματι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένωση πολιτών και θα πρέπει να μας ενδιαφέρει η ποιότητα ζωής στην Ευρώπη. Αυτό θέλω να απαντήσω και στον κύριο Γιώργ. Θα πρέπει να συνδέσουμε μεταξύ τους ε, τις διάφορες συζητήσεις που πραγματοποιούνται, διότι Έχουμε τους στόχους του κλίματος, για παράδειγμα. Εάν δεν καταφέρουμε να έχουμε ένα κοινό αφήγημα για το κλίμα, την ποιότητα του αέρα, την βιοπικιλότητα και την ε, ποιότητα ζωής, θα είναι πολύ ε, δύσκολο να γίνει κατανοητό. Νομίζω λοιπόν ότι είναι σημαντικό να συνδέσουμε μεταξύ τους τα διάφορα θέματα αυτά και να τα δούμε ως ένα σύνολο. Στον κύριο Γκερμπράντι να απαντήσω νομίζω ότι θα πρέπει να κάνω κάποιες διευκρινήσεις. Και στο άτυπο συμβούλιο και στο επίσημο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος μιλάμε για το κλίμα. Έχουμε λοιπόν ε, μια εργαλειοθήκη την οποία στέλνουμε στους Υπουργούς Οικονομικών που θα συζητήσουν το θέμα αυτό πάλι σε άτυπο και μετά σε επίσημο επίπεδο. Έχετε όμως απόλυτα δίκιο ότι θα πρέπει να ευθυγραμμίσουμε τις πολιτικές. Και δεν θα πρέπει να σκεφτόμαστε ότι πρόκειται για απομονωμένους τομείς. Θα πρέπει να έχουμε μια συνολική οπτική. Κυρία Κονέτσνα. Θέσατε κάποιες ερωτήσεις για... Αναφερθήκατε στην οδηγία για τα ανώτατα όρια εκπομπών. Και πράγματι σκοπεύουμε να προωθήσουμε το θέμα αυτό για να λυθούν τα προβλήματα και θέσατε και ερώτηση σχετικά με τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς και την προστασία των καταναλωτών. Αυτά αποτελούν αρμοδιότητα των Υπουργών Υγείας και Γεωργίας. Θα προτιμούσα λοιπόν να αφήσω αυτούς να απαντήσουν σε αυτές τις ερωτήσεις σας. Προχωρώ στις παρατηρήσεις του Μπάς Νομίζω ότι είναι πολύ φιλόδοξη η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε τον στόχο τουλάχιστον 40% και τον Σεπτέμβριο ε, θέλουμε σαφή εντολή, να είναι σαφής η πενταετής κύκλη, οι μακροπρόθεσμοι στόχοι. Ε, πρέπει να είναι σαφές ότι θέλουμε μια δυναμική συμφωνία. Θα πρέπει λοιπόν να αυξήσουμε το επίπεδο της φιλοδοξίας μας. Εάν καταφέρουμε να ξεπεράσουμε τους στόχους μας, θα είναι δυνατόν με μια τέτοια συμφωνία να έχουμε ακόμα καλύτερο αποτέλεσμα. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό όσον αφορά το κλίμα είναι να έχουμε σαφείς και κατανοητούς στόχους για όλους. Θα πρέπει να καθιερωθούν αυτοί οι μακροπρόθεσμοι στόχοι, ώστε και οι διάφοροι τομείς να προσαρμοστούν. Οι θαλάσσιοι βιότοποι αποτελούν μέρος της ε, στρατηγικής, οπότε θα εξεταστεί κατά την ενδιάμεση αναθεώρηση. Και επίσης, κύριε Ιόρκ. Νομίζω ότι ήδη ε, έχουμε στο θεματολόγιο πολλές λύσεις ε, και στο πρόγραμμα των Παρισίων. Φαίνονται, διαφαίνονται πολλές αλλαγές, ε, γι' αυτό και θα πρέπει το αφήγημά μας να αγγίξει τους Ευρωπαίους πολίτες και να συνδυάσει τις δικές μας προτεραιότητες με τις δικές τους ανησυχίες. Η πρωταρχική μας προτεραιότητα είναι η διαφύλαξη της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας. Έναν πονοπλανήτη έχουμε όλοι, συνυπάρχουμε, συμβιώνουμε σε αυτόν και περιοριζόμαστε από τα δικά του όρια. Γι' αυτό θα πρέπει να εξασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα, την αηφορία και τους τρεις άξονες της αηφορίας που είναι η οικολογία, η κοινωνία και η οικονομία. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να προβάλλουμε ώστε να έχουμε μία ενία προτεραιότητα όλοι από κοινού την διαφύλαξη της ποιότητας της ζωής των συμπολιτών μας. Ελπίζω ότι απάντησα στις περισσότερες ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ για την υποστήριξή σας. Εμείς σας ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Αυτό ήταν ο πρώτος γύρος. Περνάμε στο δεύτερο τώρα. Σίγουρα θα υποβληθούν και άλλες ερωτήσεις. Ο Μισελ Νταντά θα είναι ο πρώτος ομιλητής στο δεύτερο γύρο. Μην ξεχνάτε ότι έπεται ψηφοφορία, γι' αυτό σας θέρμα παρακαλώ να μην ξεπεράσετε το 1,5 λεπτό καθένας στο γύρο αυτό. Ο Μισελ Νταντά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Υπουργέ, καταρχήν να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στο έργο σας στα καθήκοντά σας ε, που δεν είναι καθόλου εύκολα για το επόμενο εξάμεινο. Παρουσιάστε τις προτεραιότητες σας. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσφατα ξεκίνησε δημόσιες διαβουλεύσεις για την εφαρμογή των οδηγιών για τα ιδιαιτήματα και τα πτηνά στα πλαίσια του προγράμματος ε, REFIT και θα πρέπει να αναθεωρήσει και την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Βιοπικιλότητα. Οι μελλοντικές αυτές αναθεωρήσεις και μεταρρυθμίσεις μας υποχρεώνουν να βρούμε λύσει στο πρόβλημα της των προβλημάτων στη γεωργία, ε, κυρίως ε, των θανάτων ε, ζώων από αρπακτικά, από αγρίμια και κυρίως από λύκους. Στην γεωργία είχαμε τεράστια προβλήματα και μάλιστα ο πληθυσμός των λύκων αυξάνεται τα τελευταία χρόνια. Στο, στην οδηγία για, την, για τα διατήματα ήδη έχουμε πολύ θετική αποτίμηση των αποτιμάτων, ιδιαίτερα στις αλπικές περιοχές. Ε, και η αντίδραση των ε, δημοσίων αρχών προσκρούει στην οδηγία για, το βιότοπο και τη σύμβαση της Βέρνης. Είχα την ευκαιρία να μεταβώ σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και διαρωτώ με αν το κοινωνικό μας μοντέλο είναι να βλέπουμε τους βοσκούς μας αναμένους σε πλαστικές σκηνές όπως είδα στη Ρουμανία, στην Πολωνία Στόχος μας είναι να ζουν ε, οι συμπολίτε μας σε κάποιες καλύβες όπως συμβαίνει στην Ιταλία ή στη Γαλλία, σε κάποιες περιοχές τουλάχιστον. Σίγουρα έχετε και εσείς συναντήσει ανθρώπους που έχουν υποστεί ληστεία ε, και βλέπετε πόσο ανήμποροι αισθάνονται. Φανταστείτε τι γίνεται όταν ε, ένα κοπάδι διαλύεται από ένα γρήμι. Σκεφτείτε την αδυναμία και την ε, απελπισία του βοσκού. Ε, αισθάνονται ανήμποροι και ευάλωτοι οι κτηνοτρόφοι και μερικοί έχουν φτάσει στα όρια τους ε, και δεν αντέχουν πια. Και μάλιστα στο Tour de France, αυτόν τον αγώνα ε, ποδηλάτων, ε, πολύ φοβάμαι ότι θα υπάρξουν προβλήματα τις επόμενες μέρες εξαιτίας των διαμαρτυριών των απελπισμένων κτηνοτρόφων. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ ήθελα να σας ευχαριστήσω που ήρθατε και επειδή ε, απαντήσατε για την οδηγία για τα ανώτατα όρια εκπομπών. Μήπως θα μπορούσατε να αναλύσετε περισσότερο τα πιθανά δύσκολα σημεία στο Συμβούλιο για αυτό το θέμα. Και δεύτερη ερώτησή μου αφορά κάτι που διάβασα ε, για την, προεδρία, την πρόθεση της Προεδρίας του Λουξεμβούργου να πρασινίσει το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο ενσωματώνοντας καλύτερα την ορατότητα για το περιβάλλον ε, στην οικονομική διακυβέρνηση. Μπορείτε να μας δώσετε κάποια παραδείγματα για το πώς θα προωθήσετε το πρασίνισμα της οικονομικής διακυβέρνησης της Ένωσης. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα η κυρία Γκέρλινγκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ κυρία Υπουργέ. Και εγώ θέλω να θέσω μια ερώτηση όσον αφορά την οδηγία για τα ανώτατα όρια εκπομπών. Θα είμαι σύντομη. Δεν μπορούμε να προκαταβάλουμε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας σήμερα, ούτε της ψηφοφορίας τον Οκτώβριο στην Ολομέλεια. Ε, το έχω όμως συζητήσει και γνωρίζω ότι υπάρχει κάποια έλλειψη συντονισμού με το Συμβούλιο, πράγμα το οποίο είναι λυπηρό. Αυτό που θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω είναι μπορείτε να μας διαβεβαιώσετε ότι μετά το διάλειμμα για τις διακοπές θα συζητήσετε με τον κύριο Τίμερμανς που είναι αυτός που ο τιμονιέρης πριν από αυτήν, πίσω από αυτήν την οδηγία και να εξασφαλίσετε ότι θα δεσμευθεί να προχωρήσει αυτό την υπόθεση και να δεν θα την αποσύρει. Σας ευχαριστώ. Μπέρντερ. Α, ευχαριστώ. Ναι. Ε, προσπαθούμε να σας μπερδέψουμε κάθε φορά και το πετυχαίνουμε, Πρόεδρε. Είναι ο κύριος Τόρβαλτς. Έχω μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση. Το 1953, στη διάρκεια των μεγάλων ε, πλημμυρών που έγιναν ε, καταστράφηκε ο πληθυσμός των κορμοράνων καραβοσυνένσης ε, και γι' αυτό και έγινε μια ιδιαίτερη προσπάθεια για την αποκατάσταση του είδους. Τι έγινε στη συνέχεια όμως από το 1986-87 αυτό το πτηνό μετετράπησε ε, κατάρα σε πληγή. Έχουμε πρόβλημα στη Γερμανία, στην Σουηδία, στη Δανία, στην Πολωνία, στι χώρε τη Βαλτική, πιθανότατα στο Καλίνιγκρετ, ακόμα και αν οι Ρώσοι τα αγνοούν και τα έχουμε και στη Φιλανδία. Και οι υπουργοί δεν κάνουν τίποτα. Κάθονται και τους κοιτάνε, γιατί είναι δυσάρεστη απόφαση. Θα είναι μία από αυτές τις δυσάρεστες αποφάσεις που θα πρέπει εσείς να λάβετε και περιμένω τις απαντήσεις σας. Ευχαριστώ. Thank you very much. And Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ελπίζω ότι το επόμενο εξάμεινο θα είναι επιτυχημένο. Και η ερώτησή μου αφορά δύο σημεία. Καταρχήν, κυκλική οικονομία. Η κυκλική οικονομία είναι πολύ σημαντική, ιδιαίτερα για τη γεωργία. Πιστεύετε ότι θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τους στόχους μας ε, προστατεύοντας ταυτόχρονα και τον αέρα και το έδαφος και τη θάλασσα. Επίσης, εδώ και 30 χρόνια μιλούμε για τη συγκέντρωση των ορυκτών ε, και την αξιοποίησή του στα πλαίσια τη κυκλική οικονομίας. Θα πρέπει να έχουμε και σχετικέ νομοθετικές προτάσεις όμω. Επίσης, Natura 2000. Είμαι υπέρ των στόχων του Natura 2000. Είναι θετική. Αλλά έχουμε και κάποια συγκεκριμένα σημεία εφαρμογή που θα πρέπει να προσέξουμε. Θα πρέπει να βρούμε λύσεις στα πιο επίμαχα σημεία γιατί μιλούμε για την εκτατική, εντατική μάλλον, συγγνώμη, κτηνοτροφία. Αλλά εμείς ε, έχουμε γεωργούς ε, που μετά από εκατονταετίες πρέπει να εγκαταλείψουν τα εδάφη τους. Η γεωργία δεν είναι μόνο ε, μέλισσες και λουλουδάκια. Η ασφάλεια των τροφίμων και η παραγωγή των τροφίμων είναι επίσης πολύ σημαντικά θέματα. Ο κύριος Παρνιά. Παρνιό. Ευχαριστώ κυρία, κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ κύριε Υπουργέ και ευχαριστώ και τα, και συγχαρητήριά μου για την ε, βολονταριστική πολιτική που θέλετε να ασκήσετε το επόμενο εξάμεινο. Θα το διαπιστώσουμε και την επόμενη εβδομάδα στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών του Λουξεμβούργου. Θα διαπιστώσω αυτή την πρόθεση και μαζί, γιατί θα έχω την τιμή να εκπροσωπώ τον πρόεδρο Λαβία στο άτυπο αυτό συμβούλιο. Ως ε, εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την COP21, θα ήθελα να μιλήσω για την συνεισφορά των νέων ε, μορφών χρηματοδότηση που θα είναι ο κραγωνιαίος λίθος του Πρωτοκόλου Συμφωνίας των Παρισίων τον επόμενο Δεκέμβριο. Έχουμε επιτάπητος ε, και στις συζητήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και γενικώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάποιες ε, νέους μηχανισμούς χρηματοδότησης που εξετάζονται. Για παράδειγμα, ο καθορισμός μιας σωστής ε, τιμής για τον άνθρακα για να βρούμε παγκοσμίω κατάλληλες πολιτικές για το κλίμα. Επίσης, ε, φόρος χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και ε, προσανατολισμός ενός τμήματος των εσόδων στους περιβαλλοντικούς στόχους. Επίσης, στα πλαίσια του ε, επενδυτικού προγράμματος του Juncker ε, έχουμε κάποιες περιβαλλοντικές εγγύησεις, δημόσιες επενδύσεις με οικολογικό χαρακτήρα και μεταφορά κάποιων πόρων προς το περιβαλλοντικό ταμείο. Έχουμε πολλούς χρηματοδοτικούς μηχανισμούς, πολύ ενδιαφέροντες Ερωτώ λοιπόν, από όλους αυτούς τους νέους μηχανισμούς χρηματοδότησης, ε, ποιες είναι οι προτεραιότητές σας και τι θα προβάλλετε στη συζήτηση ως προτεραιότητα. Τέλος, η γλυφοσάτη είναι ένα παραστακτόνο που χρησιμοποιείται ευρέως και ξέρω ότι το Λουξεμβούργο υιοθέτησε νομοθεσία που απαγορεύει τη χρήση της γλυφοσάτης, που είναι φυτοφάρμακο, ε, στα πάρκα και στους δημόσιους χώρους από το 2016. Θα, θα αξιοποιήσετε αυτό το εξάμεινο της Προεδρίας σας για να θέσετε επιτάπητος ε, το ζήτημα αυτό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Άουκεν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε εδώ σήμερα. Έχουμε πολλές προσδοκίες από την ε, ε, Προεδρία του Λουξεμβούργου. Εγώ θέλω να αναφερθώ στις οδηγίες Natura 2000, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές και που έχουν κάνει πολύ δημοφιλή την Ευρωπαϊκή Ένωση σε πολλές χώρες, το ότι υπάρχει δηλαδή μια κοινή στρατηγική για την προστασία της βιοπικιλότητας και για την προστασία των πτηνών. Επίσης είναι οι οδηγίες για τις οποίες έχουμε τις περισσότερες αναφορές στην Επιτροπή Αναφορών. Αυτό δείχνει πόσο απασχολεί τους πολίτες το θέμα ότι υπάρχουν οι οδηγίες αυτές και ότι έρχονται σωστά. Και στόχος δεν είναι να ξανανοίξουμε και να αποδυναμώσουμε τις οδηγίες αυτές. Και γι' αυτό ελπίζω ότι το Συμβούλιο θα προστατεύσει τους πολίτες από μια Ευρωπαϊκή Επιτροπή που σαφώς έχει δείξει ότι θεωρεί το περιβάλλον ασήμαντο πράγμα ε, στο πλαίσιο της ε, ε, πολιτικής small on small things. Ο Επίτροπος Τίμιρμανς, για παράδειγμα, ήταν πολύ ενοχλημένος που έπρεπε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης να νομοθετήσει για τις πλαστικές σακούλες. Θεώρησε ότι αυτό μπορούν να το χειριστούν ε, τα κράτη-μέλη μόνο τους. Ελπίζω λοιπόν ότι το Συμβούλιο μαζί με το Κοινοβούλιο θα προστατεύσουν τη βιοπικιλότητα στην Ευρώπη και δεν θα ξανανοίξουν τη συζήτηση για τις ε, οδηγίες αυτές. Αυτό που θα πρέπει να κάνει είναι να διασφαλίσει τη σωστή εφαρμογή τους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριο Πεντητσίνη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ που βρίσκεστε εδώ. Πρόσφατα υιοθετήσαμε μία έκθεση πρωτοβουλίας για την κυκλική οικονομία στο Κοινοβούλιο. Φαίνεται ότι το παρόν μοντέλο δεν λειτουργεί καλά και ε, κινδύνου σε για το περιβάλλον και την υγεία των πολιτών. Ελπίζουμε Λοιπόν, ε, ότι θα ε, καταλάβουμε ότι αυτό που χρειαζόμαστε είναι όχι η ανάπτυξη, αλλά η σωστή ισορροπία. Χαίρομαι που βλέπω ότι η κυκλική οικονομία αποτελεί προτεραιότητα για σας. Ωστόσο, αναρωτιέμαι Ποια κράτη-μέλη είναι διατεθειμένα να δεσμευτούν ε, για μια τέτοια πορεία. Θα πρέπει να πάρουμε σοβαρά την κυκλική οικονομία. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί η βιομηχανία μας να στηρίζεται στα παραδοσιακά όρυκτα καύσιμα. Ωστόσο, ο τομέας των ορυκτών καυσίμων έχει πολύ ισχυρό λόμπι στις Βρυξέλλες και βλέπουμε πώς επηρεάζει επίσης ε, τις αποφάσεις στα κράτη-μέλη πέρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ερώτηση λοιπόν, κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας, ε, είσαστε διατεθειμένοι να αγωνιστείτε, να καταπολεμήσετε το λόμπι του πετρελαίου ή όχι. Ευχαριστώ κύριος Φλόρενς. Κυρία Υπουργέ, Είσαστε η πεντηκοστή δεύτερη προεδρεύουσα του Συμβουλίου που συναντώ και ελπίζω ότι θα μπορέσετε με περισσότερη ενέργεια από ότι οι άντρες συνάδελφοί σας ε, να ε, ασχοληθείτε ε, με τα θέματα του περιβάλλοντος. Και θα ήθελα να πω ε, στον Γάλλο συνάδελφο ότι ε, θα οργανωθεί μία σημαντική διάσκεψη εδώ και μόνο αν έχουμε στεναρή θέση απέναντι στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο ε, θα μπορέσουμε να πετύχουμε κάτι. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μπράνεν τώρα. Σας ευχαριστώ. Δύο ερωτήσεις έχω για θέματα που δεν εξετάσαμε ακόμη. Το πρώτο φορά τη δέσμευση και αποθήκευση άθρακα, CCS, και δεύτερο βιομάζα από ξύλο. Για το πρώτο θέμα, την δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα. Από τεχνολογική άποψη, ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχετική τεχνολογία. Πρόκειται για μια τεχνολογία που απαιτεί μεγάλες επενδύσεις, αλλά θα μας βοηθήσει κατά πολέμηση των κλιματικών αλλαγών και υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξη αυτή τη τεχνολογία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποια είναι η γνώμη τη Λουξεμβουργιανή Προεδρία για τη μέθοδο αυτή, τη δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα. Και αν είστε υπέρ αυτή τη μεθόδου, πώ θα προωθήσετε το CCS στην Ευρώπη κατά το εξάμενο τη Λουξεμβουργιανή Προεδρία. Αυτή ήταν η πρώτη ερώτηση. Και η δεύτερη αφορά τη βιομάζα. Έχουμε θα αυξήσουμε την, ε, το, την καύση ξύλου, κυρίως με τη μορφή πέλετ που εισάγουμε από την Βόρεια Αμερική προκειμένου να παράγουμε ηλεκτρισμό και αυτό θα αποκτήσει μαζικές διαστάσεις. Εγώ ως Ευρωβουλευτής ε, δεν γνωρίζω αν κάτι τέτοιο είναι θετικό ή αρνητικό για το περιβάλλον. Έχουμε επιστημονικές ε, εκθέσεις που παρουσιάζουν και πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα από περιβαλλοντική άποψη αυτής της μεθόδου της καύσης ε, βιομάζας από ξύλου. Μπορείτε να μας διευκρινίσετε τις ε, περιβαλλοντικές συνέπειες ε, της μαζικής καύσης ξύλου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Πρέπει να αποτιμήσουμε περιβαλλοντικά αυτή τη μέθοδο για να δούμε τι πρέπει να πράξουμε. Τελευταίος μας ομιλητής, ομιλήτρια συγκεκριμένα, η κυρία Χέβη. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ ε, Υπουργέ, εγώ ήθελα να κάνω μια ερώτηση όσον αφορά την πρόταση αναθεώρησης του κανονισμού 1829 του 2003 για τις ε, ε, εκπομπές και την εμπορία αυτών. Θα θέσω την ερώτηση στο συνάδελφό σας το απόγευμα. Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω αυτό που μόλις ανέφερε ο συνάδελφος Παρνιό για τη χλυφοσάτη. θα έπρεπε να γίνει μια έρευνα στην οποία πιθανότατα η γλυφοζάτη θα οριστεί επισήμως ως καρκινογόνος ουσία και για το γεγονός ότι σε ορισμένα κράτη-μέλη αυτό ήδη απαγορεύεται, η χρήση του ήδη απαγορεύεται, άλλα συνεχίζεται η χρήση του. Μιλώ και για την περιοχή μου, τη Λομβαρδία, όπου γίνεται μαζική χρήση και κυρίως η παρακολούθηση, η εποπτεία, γι' αυτό είναι μια ερώτηση που θέλω να κάνω. Η ε, παρακολούθηση για αυτό το, τη χρήση αυτού του φυτοφαρμάκου ε, δεν είναι ομοιογενής. Γίνεται στη Λομβαρδία αλλά όχι στην υπόλοιπη Ιταλία. Όπως και σε άλλα κράτη-μέλη υπάρχει διαφορά ελέγχου των επιπτώσεων που μπορεί να έχουν αυτές οι ουσίες ε, για την υγεία αλλά και για το περιβάλλον. Γιατί τα στοιχεία είναι πραγματικά ανησυχητικά. Η εντατικοποίηση δε των γεωργικών πρακτικών και η χρήση φυτοφαρμάκων αλλά και λοιπασμάτων είναι ένα από τα σημαντικότερα αίτια κινδύνου για τη βιοπικιλότητα. Εάν λοιπόν σκοπεύετε να μας πείτε, ε, στο πλαίσιο της αναθεώρησης στρατηγικής για τη βιοπικιλότητα, αν σκοπεύετε μέχρι το 2020 να λάβετε σοβαρά υπόψη αυτή την πτυχή. Σας ευχαριστώ. Άλλη ερώτηση. Η κυρία Ντάλη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Υπουργέ. Ήθελα να θέσω μια ερώτηση όσον αφορά την εφαρμογή του πολιτικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την ποιότητα του αέρα, καθώς και την επίγουσα ανάγκη να, τεθεί, να δημιουργηθεί μια ε, ρύθμιση για τις εκπομπές και την ποιότητα του αέρα. Είναι ένα θέμα το οποίο εσείς αναφέρατε στις αρχικές, στην αρχική σας εισήγηση. Πώς δηλαδή θα περιοριστεί η ρήπανση του αέρα και οι εκπομπές ε, όπως ε, το μονοξίδιο του αζότου και τα μικροσωματίδια. Διαπιστώσαμε ότι υπάρχει αύξηση στις εκπομπές μεθανίου που συμβάλλουν ε, σε μεγάλο βαθμό στις γενικότερες εκπομπές. Οχήματα ευρώ, 5 και ευρώ 6 καθώς και τα βαρέα οχήματα, τα μεγάλα φορτηγά εσείς αναφέρατε, ε, αναφερθήκατε μάλλον στις οδηγίες ΕΡΟ 5 και ΕΡΟ 6 που διέπουν αυτά τα ζητήματα. Είπατε ότι αυτά βρίσκονται στις προτεραιότητες της Λουξεμβουργιανής Προεδρίας. Μπορείτε να μας δώσετε περισσότερες συγκεκριμένες λεπτομέρειες όσον αφορά το τι θα ήθελε να πετύχει η Προεδρία σας στη διάρκεια των 6 μηνών για τη βελτίωση του ποιότητας του αέρα. Πιο συγκεκριμένα δηλαδή για τις οδηγίες Ευρώ 5 και και ευρώ 6. Άκουσα πως δεν συμφωνείτε για τις κατεξουσιοδότηση πράξεις ε, συμπεριλαμβανομένου και των δοκιμών σε πραγματικές συνθήκες ε, οδήγησης όσον αφορά τις εκπομπές. αν χρειάζεται λοιπόν να διαπραγματευτούμε για να φτάσουμε σε συμφωνία ανάμεσα στο Συμβούλιο και το Ευρωκοινοβούλιο να μας ενημερώσετε. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Έχουμε ένα μέγα σύνολο ερωτήσεων και σας δίνω το λόγο ώστε να απαντήσετε σε όλα αυτά τα ερωτήματα. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσετε δε, να ολοκληρώσετε και να δώσετε τις απαντήσεις σας μέσα σε 10 λεπτά, γιατί πρέπει να ψηφίσουμε μετά. Σας ευχαριστώ πολύ. Διαπιστώνω και καταγράφω τις διεκδικήσεις του κυρίου Νταντά, το ίδιο και για τον κύριο Τόρβαλτσα σε σχέση με τα ερωτήματα του για το πράσινο εξάμεινο, το πρασίνισμα μάλλον το ε, του εξαμήνου. Είναι πολύ σημαντικό να μιλήσουμε για τις ε, επιδοτήσεις και τις σχετικές πολιτικές. Αν δείτε ότι πρόκειται για τεράστια ποσά από τα οποία ε, ε, καταλήγουν στα ορυκτά καύσιμα, ε, στα στερεά καύσιμα, αλλά και σε πρακτικές που ρηπαίνουν στην Γεωργία. Και γι' αυτό προσπαθούμε να το συζητήσουμε στη Γεωργία, γιατί όλοι γνωρίζουμε πως ε, υπάρχει πρόβλημα όταν δεν έχουμε τη σωστή ε, χρηματοδότηση. Η κυκλική οικονομία για μας είναι όντως πολύ σημαντικό θέμα, καθώς και η οικονομία ε, με επαρκή πόρους θα πρέπει να είναι και ανταγωνιστική. Γι' αυτό το λόγο και έτσι θα απαντήσω και στις ερωτήσεις του κυρίου Πετιτσίνη ότι χρειάζεται ισορροπία, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχουν τεράστια ωφέλη για την οικονομία. Ήμασταν ένα από τα 11 κρατημέλη που υπέγραψαν πέρυσι την επιστολή προς την Κομισιόν ότι δεν θα πρέπει να, να, να αποσυρθεί αυτό το πακέτο για τα απόβλητα και σκεφτόμαστε ότι θα πρέπει να διαχειριστούμε ε, σωστά τα όσα υπέβαλε ο Ποτόσνικ. Ε, Πέρσι στο Συμβούλιο 23 κατημέλη ήταν υπέρ της κυκλικής οικονομίας και υπέρ της ορθής διαχείρισης των αποβλήτων καθώς και της διατήρησης των προϊόντων στο κύκλο και στην οικονομία όσο γίνεται περισσότερο. Για μας είναι πολύ σημαντικό θέμα και θα αρχίσουμε να δουλεύουμε όσο γίνεται πιο σύντομα ε, με την κατάθεση της νέας προτάσης. Κύριε Παγνιό, ε, που είστε εισηγητής για την COP21, ε, μάλλον, για την 21. Υποβάλλατε ερωτήσεις σε σχέση με τα οικονομικά. Για μας είναι ένα στοιχείο κλειδί και ε, θέλουμε να φτιάξουμε μια εργολιοθήκη ώστε να έχουμε τη δυνατότητα ε, για όσο γίνεται περισσότερους μηχανισμούς χρηματοδότησης, νέους μηχανισμούς, ε, μέσω των οποίων θα μπορέσουμε να κάνουμε επενδύσεις, να κάνουμε πράσινη πράσινες επενδύσεις, ασφαλίσεις. Θα έχουμε τεράστιες δυνατότητες που θα βάλουμε σε ένα μια εργαλειοθήκη έτσι ώστε να αποδείξουμε ότι το οι πράσινες προτάσεις μπορούν να λειτουργήσουν. Είναι απαραίτητο να το αποδείξουμε αυτό πριν το Παρίσι για να έχουμε την εμπιστοσύνη όλων. Δηλαδή το Green Climate Fund δεν είναι το μόνο μέσο, αλλά ότι θα πρέπει να έχουμε διάφορα μέσα για να μπορέσουμε να πετύχουμε διάφορα πράγματα, εφόσον μιλάμε για κλιματική χρηματοδότηση και να έχουμε και τη δυνατότητα να προχωρήσουμε στα 100 δις ετησίως από το 2020, ότι θα είναι κάτι τέτοιο εφικτό και ότι η Ευρώπη θα παίξει τον υπηκοδομητικό της ρόλο στη συζήτηση αυτή. Για την ε, γλυφοζάτη, σάτη, με συγχωρείτε, Είναι μια τεράστια πρόσκληση, πρόκληση. Πρέπει να όμως να συνεργαστούμε σε διεθνές επίπεδο. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα. Η κυρία Όκεν, βιοπικιλότητα, ευχαριστώ για τη δήλωσή σας και συμφωνώ. Και ελπίζω προσβλέπω στην συνεργασία σας, στη σύρρηξή σας για αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ. ευχαριστώ επίσης τον κύριο Φλόρενς για την παρέμβασή του. Η εφαρμογή πράγματι είναι αποφασιστικής σημασίας. Πέρα από την εφαρμογή όμως θα πρέπει να λαμβάνουμε πάντα υπόψη και την χρηματοδότηση. Και εδώ ακριβώς έχουμε το θέμα της ευθυγράμμισης των πολιτικών. Κύριε Μπράνεν. Όσον αφορά το σύστημα εμπορίας εκπομπών, ε, Όσον αφορά την δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα, αυτό ε, θα γίνει σήμερα μία συνάντηση γενικών διευθυντών και νομίζω ότι περισσότερο πρέπει να μιλήσουμε για την ευθυγράμμιση των πολιτικών. Θα πρέπει να πούμε ότι χρειαζόμαστε μία βιώσιμη προσέγγιση όσον αφορά την αλλαγή του κλίματος. Κυρία Ελενοριαίδη. Το θέμα της ε, γλυφοσάτης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να παρακολουθήσουμε την κατάσταση. Περιμένουμε τα αποτελέσματα της μελέτης ε, και πρέπει να μιλήσουμε όχι μόνο για τη γλυφοσάτη, αλλά και για την χρήση των φυτοφαρμάκων γενικά. Και τέλος, όσον αφορά την ποιότητα του αέρα και το κλίμα. Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και είμαστε διατεθειμένοι να συνεργαστούμε με το Κοινοβούλιο και να πετύχουμε πολιτική συμφωνία. Γνωρίζουμε ότι θα είναι δύσκολο αυτό, κάνουμε όμως ό,τι μπορούμε. Και νομίζω ότι ξέχασα την κυρία Γκέρλινγκ. Ήθελα να σας πω ότι πρόσφατα είχα επαφές με τον Γενικό Γραμματέα σχετικά με την ερώτησή σας. Είχα πρόσφατα επαφές και Μιλήσαμε ακριβώς για το θέμα αυτό. Είμαστε πεπισμένοι ότι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε, θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια όσον αφορά τα θέματα ποιότητας του αέρα και τα εθνικά όρια εκπομπών. Thank Πάθησα να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις. Σας ευχαριστούμε θερμά κύριε Υπουργέ. Μπορούμε να ολοκληρώσουμε αυτό το πρώτο τμήμα της ε, συνεδρίασής μας. Ευχαριστούμε την Υπουργό Περιβάλλοντος του Λουξεμβούργου για την πολύ χρήσιμη αυτή ανταλλαγή απόψεων που είχαμε και για την ευκαιρία που μας δώσατε ε, να γίνει συζήτηση και που την προθυμία να απαντήσετε σε όλες αυτές τις ερωτήσεις. Μία πολύ σύντομη διακοπή για να περάσουμε στις ψηφοφορίες.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 Okay, it uh, time to start Να ξεκινήσουμε τις ψηφοφορίες. Πρέπει πρώτα όμως να κάνω μια ανακοίνωση. Ο Μάρτιν Φούξ θα αποχωρήσει από τη γραμματεία μας και θα πάει στην γραμματεία της Επιτροπής Τραν. Θέλω τον ευχαριστήσω για την υποστήριξή του προς ε, τα μέλη της ΕΝΒΗ. Και να του ευχηθώ καλή επιτυχία στη νέα του θέση. και μπορούμε να ξεκινήσουμε με το θέμα υπαριθμών 5 της ημερήσιας διάταξης που είναι ε, ο περιορισμός των εκπομπών ορισμένων ρήπων στην ατμόσφαιρα από μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης. Μπορούμε να προχωρήσουμε κατευθείαν στην ψηφοφορία. Αρχή της ψηφοφορίας. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε. Have you voted? Ψήφισατε παρακαλώ. Λήξη της ψηφοφορίας εγκρίθηκε. Και μπορούμε τώρα να προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα της ημερησίας διάταξής μας. ψηφίζουμε την επόμενη οδηγία. Να συγχαρούμε τον εισηγητή, τον κύριο Γκζιπ και προχωράμε στην ψηφοφορία. της επόμενης έκθεσης που έχει πολύ ογκώδη κατάλογο ψηφοφορίας είναι η έκθεση της κυρίας Γκέρλινγκ, τροπολογία 14α της Επιτροπής Άγκρη. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Check. Sorry. Να ελέγξουμε ένα λεπτό. Avete Ψηφίσατε όλοι. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Α, λυπούμε. Ωραία, ξεκινάμε. Τροπολογία, μάλλον υπήρξε μια καθυστέρηση με τη μετάφραση. Ε, περιπτώσει. Τροπολογία 127. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5 ως προσθήκη στη συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε την τροπολογία ΙΤΡΕ 9 ίδια με την 128 και 129 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τώρα ψηφίζουμε την συμβαστική 4α. Τέσσερα. Έχω κάποιες λαθάκια στο κατάλογο ψηφοφοριών μου. Συμβιβαστική 4. α τεσσερα εχω καποιες και στο καταλογο ψηφοφοριων μου συμβιβαστικη 4 λοιπον ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκαινέται. Συμβαστική 22 καταπίπτει και ψηφίζουμε την συμβαστική 4α. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 155. Έκαουτ και άλλοι. Υπέρ. Κατά. Αποχές έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι, τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 18 τώρα. υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 19 τώρα, υπέρ. Κατά, αποχές, έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι, τέλος ψηφοφορίας, εγκρίνεται. Page 16, compromise 21. Dobbiamo votare adesso il compromesso. Τώρα πρέπει να ψηφίσουμε τη συμβιβαστική 21. Σας δίνω το χρόνο να το βρείτε γιατί κάναμε μέγα άλμα στον κατάλογο ψηφοφορίας. Συμβιβαστική 21. Compromesso 21. Chi è a Συμβαστική 21 λοιπόν. Ποιοι είναι υπέρ, κατά. εποχέ. Εγκρίνεται. Αλλά α, θα κάνουμε και έναν ηλεκτρονικό έλεγχο. Ψηφίσατε όλοι. Εγκρίθηκε. Votiamo adesso L'emendamento ITRE 312 i 12, τροπολογία e i Η312. E e Emendamento ITRE Η312. Chi è a favore? Τροπολογία Ήτρε 12. Ποιοι είναι υπέρ κατά εμποχές, απορρίπτεται. 16 το εισηγητή. Υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. 183 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 184 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος. Έχουμε έναν παραπάνω από το ΕΛΚ. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τώρα την τροπολογία Άγκρη 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 186 υπέρ, κατά, εποχές απορρίπτεται. Καλά, του χρόνου τέτοια μέρα. Ε, ψηφίζουμε τώρα την 187 γιατί η συμβιβαστική 22 δεν εγκρίθηκε. 187 λοιπόν τώρα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ήτρε 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική μάλλον ε, ένα ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία ποιετικά είναι υπαριθμών 209. Ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 212. Κονέτσνα, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 215, γιατί 22 δεν εγκρίθηκε. 215, υπέρ, κατά, αποχές έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Ε, απορρίπτεται. Τροπολογία 213 μέχρι 214. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, εγκρίνονται. Τροπολογία 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 216. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ήτρε 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές ε, ε, απορρίπτεται. Ήτρε 17. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 217 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 232 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία Ήτρε 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 222 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογίες 22, 228 είναι ταυτόσιμες, ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται. 219 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογίες 220 και 221 που είναι ταυτόσιμες, ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Απορρίπτονται. Τροπολογία 23 της εισηγήτριας, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία Ήτρε 18 υπέρ, κατά. Ήτρα 18, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 24, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 228, Μπέρντερ και Φέντερλε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 229 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 230 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ε, έλεγχος, εντάξει. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 231. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα ψηφίζουμε τη συμβιβαστική 15. Συμβιβαστική 15 ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα ψηφίζουμε την τροπολογία 251 των Καπούτο και άλλων. Ε, Υπέρα ποιοι είναι κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 252 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος πληροφορία Εγκρίνεται. 254. 254. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 257. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ταυτόσιμες τροπολογίες 261 και 320. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται. Ψηφίζουμε τις τροπολογίες την τροπολογία 259. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 260. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 262 και 263 ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται απορρίπτονται τροπολογία 264 ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 5 υπέρ Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Votiamo adesso l'emendamento 260. Τροπολογία 269 της συναδέλφου Κονέτσνα. Ποιοι είναι υπέρ. Chi è contro? Chi si astiene? Κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογίες 270, 271, 272, 73 και 321 που είναι ταυτόσιμες. Υπέρ ποιοι είναι, κατά, αποχές, απορρίπτονται. 274. Βυσνιεύσκα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 275 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία Ήτρε 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογίες 276-277 που είναι ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τώρα ψηφίζουμε την τροπολογία 278. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 279. Ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Και τώρα ψηφίζουμε την συμβιβαστική 3. Συμβιβαστική 3 ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Votiamo adesso il... Votiamo adesso il compromesso 16. Συμβαστική 16 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογίες ταυτόσημε. 293 και 294. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. Άγκρι 31. Ε, Ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Dobbiamo votare adesso l'emendamento 297. 297 τώρα. Τροπολογία 297, ποιοι είναι υπέρ. Chi è contro, chi si astiene, respinge. Αποχές απορρίπτεται. 298 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 291-301-302 υπέρ. Κατά αποχές έλεγχος. Avete votato tutti, il voto è Ψηφίσατε όλοι, απορρίπτονται. Για μια ψήφο. Τώρα ψηφίζουμε την τροπολογία 300. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 305. 305. Τρακόσια ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία άγκρι 33. Άγκρι 33, ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές, έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Αγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα τη συμβιβαστική 17 υπέρ. κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ κατά Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική υπαριθμών 6. Υπέρ. Α, όχι, όχι. Πρέπει να ψηφίσουμε την άγκρη 36 πρώτα. Υπέρ. Άγκρη 36. Κατά. Α, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα ψηφίζουμε την τροπολογία 348 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 350 υπέρ αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 352 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 24 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την τροπολογία ΙΤΡΕ 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ταυτόσημες 358 και άγκρι 38. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τώρα ψηφίζουμε τη συμβιβαστική 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και τώρα περνάμε στην τροπολογία 46 της εισηγήτριας, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 362, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 363. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 364 και 365 και 66 που είναι ταυτόσιμες με την Ήτρα 34. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Απορρίπτονται. Ήτρα 35. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 6. Ταυτόση με την άγκρη 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7 της εισηγήτριας υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Άγκρη 18 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 8 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα την τροπολογία 11 της εισηγήτριας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 134 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. Τροπολογία 136. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παρακαλώ να ζητήσω από τους σοσιαλιστές να σηκώνετε τα χέρια σας. Ψηφίζουμε τώρα για την τροπολογία 137. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία Gzib. 367 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 362 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 363 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 412 412 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 413 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Θέλετε έλεγχο. Οκ. Okay. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 414. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Άγκρι 44 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 415 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 45, άγκρι 45, ε, ποιοι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 417, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 418, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 419 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Ήτρε 41 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Τροπολογία 420 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Συμβιβαστική 9 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 10 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Αγκρι 48 ε, τώρα. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 427. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 428 και 429 είναι ταυτόσιμες, τις ψηφίζουμε υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 430 και 431. Υπέρα. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 432 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Avete votato Ψηφίσατε όλοι. Τέλος της ψηφοφορίας απορρίπτεται. 433. 433 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 434 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 435 και 436 είναι ταυτόσιμες υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται. Επειδή η συμβαστική 23 δεν ψηφίστηκε, πρέπει να ψηφίσουμε το 437 και 441 ε, ε, υπέρ. Κατά. Οι σοσιαλιστές τι ψηφίζετε. Κανένας δεν σήκωσε το χεράκι του. Έλεγχος ηλεκτρονικός. Avete votato tutti? Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται 438 και 439 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ήτρε 42 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 440 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογίες 442 και 443 που είναι ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 444 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 445 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 446 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 447 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 448 και 449 είναι ταυτόσημες. Υπέρ ποιοι είναι. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 451 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 452 453, 454. Είναι ταυτόσιμες ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 456 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 458 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 459. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 460. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 461 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 464, 465 ε, που είναι ταυτόσημες. Υπέρ ποιοι είναι. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 469 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 468 ε, υπέρ. 468 υπέρ. Κατά. Αποχές έλεγχος. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Ψηφίσατε όλοι, απορρίπτεται. Ψηφίζουμε την 470. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τετρακόσια εβδομήντα ένα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 474. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 472, 473 πανομοιότυπες. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Ψηφίζουμε τώρα την 475. Ποιος είναι υπέρ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τις τροπολογίες 476, 477 και 478. Ταυτόσιμες. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Ψηφίζουμε τη συμβαστική τροπολογία 12. Ποιος είναι υπέρ. Υπέρ της συμβαστικής τροπολογίας 12. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε στη στην τροπολογία 483. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ψηφίζουμε την 484 του κυρίου Φλόρεντς. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 485. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 486. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 487. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 488. ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 489 και άγκρι 50 που είναι πανομοιότυπες. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνονται. 493 τώρα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 494. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 11. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 50. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 501 που είναι πανομοιότυπη 502; Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 517. Τζέσικα και Πέτερ Γιάρ. Ποιος είναι υπέρ της 517. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε την 518. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 519 και Ήτρε 43. Πανομοιότυπες. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος. Avete votato tutti, il voto è chiuso. όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτονται. 520. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 521. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Αιτιολογικές σκέψεις. 52. Τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 54. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 56. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 57. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Άγκρι 2. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 58. Τροπολογία ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίζετε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Ήτρε 2. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 60. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 67. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 63 και 64 ταυτόσημες. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 65. Ποιος είναι υπέρ. Υπέρ της 65. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 66 και άγκρι 4. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. Τροπολογίες 68 και άγκρι, 5 που είναι πανομοιότυπες. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι, τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτονται με μία ψηφοδιαφορά. Ψηφίζουμε την τροπολογία Άγκρι 3. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές Απορρίπτεται. Τροπολογία Ήτρε, υπαριθμό 5. Ποιος είναι υπέρ της πέμπτης τροπολογίας της Επιτροπής Ήτρε. Κατά. Οχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 78. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Άγκρι 7. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 79. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 80. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 82. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 81. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 83. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Μια και η 89 τροπολογία έχει εγκριθεί, Τροπολογίε 85 σε 86 β ε, και 87 β καταπίπτουν. 92 α τώρα, Ποιο είναι υπέρ, Ποιο είναι υπέρ, επαναλαμβάνει ο πρόεδρο. κατά αποχές απορρίπτεται. Προχωράμε. Κατέπεσαν οι ενδιάμεσες τροπολογίες. Περνάμε στην 101. Ντάν Καπούτο, ε, Μπραντλάιν και Μπροκ. Ψηφίζουμε την τροπολογία 101. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Avete Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 108. οκτώ. Εκχάουτ, Πεντιτσίνη και Λυπή. Ποιος είναι υπέρ της 108. Κατά. Εγκρίνεται. 112. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 109 και 110 ταυτόσημες ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 111 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 113 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 114 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 117 ποιος είναι υπέρ υπέρ της 117 κατά αποχές εγκρίνεται 118 ποιος είναι υπέρ Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 118. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Άγκρι 12. Ποιος είναι υπέρ της τραπολογίας 12 της Επιτροπής ε, Γεωργίας κατά αποχές απορρίπτεται 122 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Ήτρε 8 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Ψηφίζουμε την στραποποιήθησα πρόταση ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Λήξη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και το νομοθετικό ψήφισμα τώρα, ηλεκτρονικά και πάλι, άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Και τώρα πρέπει να ψηφίσουμε τις τελευταίες, την τελευταία έκθεση για σήμερα. If Αν είστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε, πρόκειται για την έκθεση για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την περιοχή της Αιδετικής και του Ιωνίου. Ο εισηγητής είναι ο κύριος Αφρόντε. Συμβιβαστική ένα. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τώρα ψηφίζουμε την τροπολογία 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 12. Υπέρ. Κατά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 Τροπολογία 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 20, 30 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 31 υπέρ κατά έλεγχος. Avete votato Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Ε, απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τώρα την τροπολογία 34. Ποιοι είναι Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Ε, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 40. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ε, τροπολογία 47. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είδα. Τροπολογία 47. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 50. Ε, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 5. Υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 58 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 59 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται.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 το σχέδιο γνωμοδότησης όπως τροποποιήθηκε. Ποιοι είναι, ε, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ το συνάδελφο Αφρόντε. Ολοκληρώθηκαν έτσι οι ψηφοφορίες. Ε, Δύο λεπτά διάλειμμα και μετά ξαναρχίζουμε όταν ε, όσοι δεν ενδιαφέρονται για τη συνέχεια θα έχουν φύγει από την αίθουσα.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 Αγαπητοί συνάδελφοι, μπορούμε να προχωρήσουμε στο σημείο 9 της ημερησίας διάταξης. Πρόκειται για εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης για τον Γενικό Προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016. Και θα ξεκινήσουμε δίνοντας το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ακούσουμε τις θέσεις της Επιτροπής και να μας ε, κάνει την παρουσίασή της. Δίνω το λόγο λοιπόν κατευθείαν ε, στη Φρανσουάς Καζάνα ή Λεκλέρκ. Παρακαλώ, ξεκινήστε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Λέγομαι Ντεκλέρκ και εκπροσωπώ την Γενική Διεύθυνση ε, Ασφάλειας Τροφίμων. Έχουμε λοιπόν δύο προγράμματα. Έχουμε το πρόγραμμα υγείας και των τροφίμων και ζωοτροφών για το 2016. Πρόκειται για το τρίτο έτος του σε δημοσιονομικού πλαισίου και όσον αφορά τις αναλήψεις υποχρεώσεων δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Όσον αφορά τις ε, πληρωμές όμως, ε, το 2014 δεν είχαμε κανένα πρόβλημα με το πρόβλημα δημόσιας υγείας, ούτε περιμένουμε προβλήματα μέχρι το τέλος αυτού του έτους, ούτε του επόμενου. Όσον αφορά το πρόγραμμα τροφίμων και ζωοτροφών, μια επιστροφή προς κράτος μέλος δεν ε, μπόρεσε να γίνει μέχρι το 2014, έγινε μόνο εν μέρη, πληρώθηκε αρχές του 2015. Δεν περιμένουμε να υπάρξει κανένα συγκεκριμένο πρόβλημα μέχρι το τέλος ε, αυτής της χρονιάς ε, και το ποσό που έχει διατεθεί για τις πληρωμές το 2016 επίσης θα πρέπει να θεωρηθεί επαρκές. Η γενική μας διεύθυνση είναι επίσης αρμόδια για αποκεντρωμένους οργανισμούς. Έχουμε την CPVO που χρηματοδοτείται αποκλειστικά από τα τέλη. Μετά έχουμε δύο που εν μέρη χρηματοδοτούνται έτσι, η ΕΜΑ και οι ε, δραστηριότητες για τα βιοκτώνα της ΕΑ. Ε, και μετά έχουμε την ΕΦΣΑ και την ECDC που εξαρτώνται αποκλειστικά από δική μας χρηματοδότηση. Το προσωπικό τεσσάρων ε, από αυτούς τους οργανισμούς ε, ε, ανταποκρίνεται απολύτως στην σχετική έκθεση της Κομισιόν το 2013 για την ΕΚΑ. Υπάρχει ε, διαφορετική ρύθμιση διότι αναμένεται ότι θα πρέπει να αναθεωρηθεί το ποσό της ενίσχυσης όπως επίσης και το μέγεθος του προσωπικού όσον αφορά τα πιλωτικά προγράμματα και τις προπαρασκευαστικές δράσεις. Έχει σταλεί έκθεση στο Κοινοβούλιο. Έχουμε έγγραφα εργασία σε το μέρος 4 ε, του Ιουνίου του 2015, όπου αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες για τα πιλωτικά προγράμματα. Δεν έχουμε παρατηρήσεις για τη γνωμοδότηση. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Ευχαριστώ. Λέγομαι Φρανσουά Καζανά, Διπροσωπεύω την Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Κλιματικής Δράσης. Έχουμε ένα πρόγραμμα, το LIFE, που αφορά αυτές τις δύο γενικές διευθύνσεις, εν τέταρτο της γάμα δέλτα κλίμα και τρία τέταρτα γάμα δέλτα περιβάλλον. Ε, το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2016 ε, στο ισχύον οικονομικό πλαίσιο. Χαρακτηρίζεται από αύξηση κατά 6,4% των πιστώσεων ανάληψη υποχρεώσεων, όπως πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οπότε έτσι θεωρώ ότι θα καλύψουμε τις νέες μας ε, δεσμεύσεις σε ό,τι αφορά τα προσχρηματοδότηση προγράμματα και σχέδια για το 2016. Όπως ξέρετε, ένα τμήμα του προγράμματος, η διαχείριση ενός τμήματος του προγράμματος ανατέθηκε σε μια εκτελεστική υπηρεσία, σε ένα εκτελεστικό οργανισμό που θα διαχειριστεί όλα τα νέα προγράμματα και η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος θα συνεχίσει να διαχειρίζεται τα παλιά προγράμματα, τα παλιά σχέδια που εκείνη είχε ξεκινήσει και που γνωρίζει καλά. Έχουμε και τον οργανισμό της Κοπενχάγης, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος δηλαδή. Οι προτάσεις γι' αυτόν βρίσκονται στην ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έχουμε και μια συγκεκριμένη δημοσιονομική γραμμή που αφορά τις πολυμερείς συμφωνίες και τις διεθνείς συμβάσεις. Εκεί ζητούμε αύξηση της αντίστοιχης δημοσιονομικής γραμμής γιατί θα έχουμε και νέες συνεισφορές για τη βιοπικιλότητα και με τις συμφωνίες της Ναγκόγια και το πρωτόκολλο ΣΥΤΕΣ. εξαιτίας της προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια νέα σύμβαση για τα διασυνοριακά χωρικά είδατα. Είναι αρκετά λεπτό αυτό το θέμα της ε, σχετικής δημοσιονομικής γραμμής γιατί εξαρτάται πολύ από την ε, ισοτιμία του ευρώ σε σχέση με το δολάριο γιατί πολλά κονδύλια καταβάλλονται σε δολάρια. Και το αρχικό αίτημα ε, κλαδεύτηκε από το Κορεπέρ, ε, περικόπηκε από το Συμβούλιο, οπότε έχουμε κάποιες ανησυχίες για τις σχετικές δημοσιονομικές γραμμές για το 2016. Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των πληρωμών, Είμαστε φέτος πιο αισιόδοξοι από πέρυσι ε, για το 2015 γιατί τα ποσά φαίνεται ότι θα μας επιτρέψουν να επιστρέψουμε σε μια ομαλότητα ε, το 2016 ε, για τις πιστώσεις πληρωμών σε σχέση με, τα, με τις ανάγκες. Και αυτό οφείλεται στο γεγονό ότι πολλοί δικαιούχοι δεν έχουν ακόμη υποβάλει τις αιτήσει πληρωμών. Οπότε θα αναβληθούν για το τέλος του έτους ή τις αρχές του επόμενου έτους. Οπότε περισσότερους δικαιούχους οφείλεται η θετική κατάσταση παρά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πάντως θεωρούμε ότι οι πληρωμές την επόμενη διετία θα μπουν σε καλύτερο δρόμο από ό,τι ήταν πέρυσι. Αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τώρα ως υπεύθυνο για τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος θα προβώ και εγώ σε κάποιους προβληματισμούς όσον αφορά τον προϋπολογισμό. Η Επιτροπή είναι πεπισμένη ότι το υψηλός βαθμός προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας εντός της Ένωσης είναι μια ε, προϋπόθεση οκτανών κάνεφε για την ε, οικονομική ευημερία και ότι η ασφάλεια των τροφίμων αλλά και των ζωοτροφών καθώς και τα όσα ο άνθρωπος προκαλεί με προξενεί μάλλον τις φυσικές καταστροφές είναι πράγματα τα οποία πρέπει να παρεμποδιστούν. Άρα λοιπόν οι γραμμές που συνδέονται με τα λίγα προγράμματα που στηρίζουν αυτούς τους στόχους θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν σωστά και μια περικοπή σε αυτές τις γραμμές δεν θα ήταν ανεκτή για μας. Από την άλλη πλευρά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η προστιθέμενη αξία των ευρωπαϊκών πολιτικών για τις πολιτικέ περιβάλλοντο είναι, είναι υψηλή και ότι τέτοιε γραμμέ έχουν αντίκτυπο πολύ θετικό για το περιβάλλον αλλά και για την ανθρώπινη υγεία τα συνολικά κονδύλια όσον αφορά τις υποχρεώσεις και τις πληρωμές ε, είναι σύμφωνες με το προϋπολογισμό και τους πόρους που προβλέπονται στο πολιετές ε, πλαίσιο για το 2016. Αλλά όπως έγινε και σε προηγούμενα έτη, υπάρχει αρκετά μεγάλη ε, ε, ανησυχία όσον αφορά το, σε καθυστερήσεις πληρωμών, γιατί η Κομισιόν γνωρίζει πολύ καλά ότι ήδη εδώ και κάποια χρόνια, στο τέλη του χρόνου, βρεθήκαμε με πληρωμές παραπανίσχες που έπρεπε να καταβληθούν σε σχέση με τη δυνατότητα ή την... Α, ε, έλλειψη βούλησης από πλευράς του Συμβουλίου να καλύψει αυτές τις δαπάνες. Αυτές μεταφέρνονται διαδοχικά στα επόμενα χρόνια. Ε, και όσον αφορά λοιπόν τις πληρωμές και τις αποζημιώσεις των κρατών μελών για τις ε, ε, προκαταβολές αυτό δεν είναι πρόβλημα αλλά για πολλά προγράμματα καθυστέρηση των πληρωμών σημαίνει και καθυστέρηση και των προγραμμάτων και αυτό το είδαμε στα προηγούμενα χρόνια και βλέπουμε και τον αντίκτυπο στα προγράμματά μας. Τώρα για το LIFE. Η Κομισιόν ε, δέχεται την, 20, την αύξηση κατά 27,7 εκατομμύρια ε, το προϋπολογισμό αυτού του προγράμματος. Όμως αυτό αποτελεί μόνο το 0,3% του συνόλου των προγραμμάτων και του σχεδίου προϋπολογισμού του για το 2016 και μόνο ε, ένα ελάχιστο ποσοστό στον τίτλο 2 και ότι ένα τέτοιο ποσοστό, αν και είναι θετικές οι επιπτώσεις για το πρόγραμμα LIFE, έχουν μείνει σταθερές εδώ και πολλά χρόνια. Για τις υπόλοιπες γραμμές του προϋπολογισμού υπάρχουν, ε, εξακολουθούν να υπάρχουν κάποιες ανάγκες για αναβολή τον ε, ε, μεταφορά μάλλον των κονδυλίων ε, υποχρεώσεων και πληρωμών με βάση τα όσα ισχύουν για το πολιτές πλαίσιο, αλλά δεν μπορούμε παρά να αναφέρουμε τις ανάγκες των οργανισμών. Στο σχέδιο προϋπολογισμού που μόλις συστάθηκε, ορισμένοι οργανισμοί μπαίνουν στο καλάθι των εξοικονομήσεων, ιδιαίτερα όσον αφορά το προσωπικό τους. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ορίσει έναν στόχο για το, για το πολιετές πρόγραμμα και αυτό επηρεάζει και τους οργανισμούς ε, όσον αφορά τη μείωση και την περικοπή του προσωπικού και όπως ξέρετε οι οργανισμοί, η ΕΜΑ και η ΕΚΑ συγκεκριμένα έχουν ε, ε, επιπλέον προϋπολογισμό που προέρχεται από τα έσοδα των ίδιων των οργανισμών λόγω των ε, παροχών που προσφέρουν. Η ΕΜΑ κυρίως αλλά και η ΕΚΑ μετά από τα όσα κάνουν για τα βιο κτώνα βρίσκονται σε μεγάλες δυσκολίες γιατί αφού από τη μια πλευρά τους αναθέτουμε επιπλέον καθήκοντα αλλά από την άλλη όμως περικόπτουμε τις θέσεις που έχουν στη διάθεσή τους το προσωπικό που έχουν στη διάθεσή τους για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις δεσμεύσεις που τους αναθέτουμε ε, Άρα λοιπόν, και ως προς αυτό θα ήθελα να ζητήσω από την Κομισιόνα να προσέξει ιδιαίτερα, γιατί δεν θα θέλαμε να ανατεθούν νέα καθήκοντα, που όμως δεν θα μπορούν να υλοποιηθούν λόγω της έλλειψης του απαραίτητου προσωπικού. Και πριν να ολοκληρώσω θα κάνω και μια αναφορά στα πιλωτικά προγράμματα και στις προπαρασκευαστικές δράσεις. Σήμερα έχουμε μια συνάντηση με τον Γενικό Συγητή του Προπολογισμού Ζωζέ Μανουέλ Φερνάντε και με όλου του συγητέ για τον Προπολογισμό 2016 για να συζητήσουμε και για τι προτεραιότητε και τα πιλωτικά προγράμματα για τα οποία λάβαμε την ε, πρώτη εκτίμηση από πλευρά τη Κομισιόν χθες ή προχτές. Από, τα 23 προτάσει που στείλαμε Εμεί από την Επιτροπή ΕΜΒΗ, μία δεν αξιολογήθηκε γιατί υπήρχε σε ένα πρόγραμμα το οποίο αυτή τη στιγμή εφαρμόζεται, ενώ οι υπόλοιπε ε, έγιναν 15 εκτιμήσεις C, 3D, 3Β και μόνο μία Α. Δηλαδή ένα πιλωτικό πρόγραμμα το οποίο πρέπει να, μπορεί να εφαρμοστεί όπως υποβλήθηκε. Είναι σαφές λοιπόν και επαναλαμβάνω και στους συναδέλφους να αναδιατυπώσουν τα πιλωτικά προγράμματα σε συμφωνία με τις συστάσεις έτσι ώστε μεγαλύτερος αριθμός πιλωτικών προγραμμάτων να είναι εφαρμοστέα, εφαρμόσιμα και άρα να μπορούν να μπουν στην τελική συμφωνία ε, που θα γίνει στην ε, Επιτροπή Προϋπολογισμού. Και γι' αυτό καλώ όλους τους συναδέλφους να ε, προσέξουν πολύ σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ και θέλω να δώσω το λόγο στον κύριο Γκρότε, αμέσω που το ζήτησε. Ευχαριστώ πολύ. Μιλώ εκ μέρους της συναδέρφου Κάριν Κάντεμπαχ που δεν μπορεί να είναι παρούσα σήμερα. Είναι μόνιμη εισηγήτρια για την πολιτική μας ομάδα όσον αφορά τα θέματα προϋπολογισμού και μου ζήτησε να πω ότι επικροτεί την γνωμοδότηση του συναδέρφου Λαβία που είναι η συγητής μας. Όλοι οι τομείς έχουν καλυφθεί επαρκώς. όσον αφορά το LIFE, τα πιλωτικά προγράμματα, το Horizon 2020, η έρευνα, όλα αυτά έχουν συμπεριληφθεί. Έχουμε το πρόβλημα των αποκεντρωμένων οργανισμών και η Καριν Κάντενπαχ επισημαίνει ότι υπάρχει εδώ μια ιδιαιτερότητα. Ο συνάδελφος Λαβία αναφέρθηκε στο προσωπικό των οργανισμών αυτών. Ε, άλλωστε, ο συνάδελφος επεσήμανε ότι χρηματοδοτούνται μέσω των τελών. Ε πληρώνουν τέλη, άρα είναι πελάτες και γι' αυτό θα πρέπει και οι ε, οι υπηρεσίες να παρέχονται σε επαρκές χρονικό διάστημα. Έχουμε πελάτες εδώ, δεν μπορούμε απλά δηλαδή να μειώσουμε το προσωπικό. Συμφωνούμε λοιπόν με τον ε, συνάδελφο Λαβία. Η Κάριν Κάντενπαχ θα υποβάλει δύο σημαντικές τροπολογίες. Η μία έχει να κάνει με το, τη χρηματοδότηση του προγράμματος για τις ανισότητες ε, στην υγεία και η άλλη ε, θα έχει να κάνει με την γεωργία, την φιλική προς το περιβάλλον, θα υποβάλει λοιπόν δύο τροπολογίες. Ε, νομίζω όμως ότι έχει δώσει πολύ καλό βαθμό ε, στον συνάδελφο Λαβία που είναι και πρόεδρος και εισηγητής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Ματίας. Δίνω το λόγο στην κυρία Κονέτσνα. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρότασή σας και νομίζω ότι ε, περιλαμβάνει πολλά από τα σημεία που επισημάναμε κατά την έναρξη της συζήτησης για το υπροπολογισμό. Ε, δεν μπορώ όμως να είμαι ικανοποιημένη για ε, με το, τη χρηματοδότηση του ECDC για την επόμενη χρονιά, διότι θα πρέπει να μετακομίσει, χρειάζεται νέα έδρα και πέρσι ε, αναθέσαμε πολλά νέα καθήκοντα στην υπηρεσία αυτή ε, που συνδέονται με τον έμπολα και άλλες μεταδοτικές ασθένειες ε, στην Ευρώπη που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία του κόσμου. Και νομίζω ότι η μείωση του προϋπολογισμού δεν θα έχει θετικές επιπτώσεις. Δεν πρόκειται για οργανισμό ε, που να σπαταλάει τους ανθρώπινους πόρους του. Ε, οι εμπειρογνώμονες και το προσωπικό μόλις που αρκούν για να ανταποκριθούν ε, στα καθήκοντα που τους αναθέτουμε. Είναι λοιπόν λανθασμένη η απόφαση για οποιαδήποτε περικοπή. Θα υποβάλω σχετική τροπολογία, διότι δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό ως πρόσωπο επαφής με αυτόν τον οργανισμό. Νομίζω ότι κάθε ευρώ που επενδύεται σε αυτόν τον οργανισμό είναι ευρώ που επενδύεται στην υγεία και την ασφάλεια των πολιτών μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος Γιάβορ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να συμφωνήσω με τους συναδέλφους. Πιστεύω ότι το σχέδιο έκθεσης του Προέδρου μας αποτελεί πολύ καλή σύνοψη της προοπτικής της ΕΝΒΗ για τον προϋπολογισμό του 2016. Θα ήθελα να προσθέσω δύο πράγματα σε αυτά που ήδη αναφέρθηκαν. Πρώτον, όσον αφορά τους οργανισμούς, θα ήθελα να τονίσω τον ρόλο της ΕΦΣΑ. Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, ε, πιστεύω ότι στην ΕΦΣΑ θα ε, επιβληθεί επιπλέον ε, φόρτος εργασίας τα επόμενα χρόνια και είναι απαράδεκτο να μην διασφαλίσουμε τους απαραίτητους πόρους για να μπορεί η ΕΦΣΑ να εργάζεται με τρόπο σωστό. για να ανταποκριθεί στον, στη διαδικασία αδειοδότηση των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Η ΕΦΣΑ λοιπόν είναι πολύ σημαντικό θέμα και όσον αφορά το LIFE ε, και ε, το πρόγραμμα για την ε, φύση, για τη διατήρηση της φύσης. Οι βελτιώσεις που έχουν υπάρξει στο περιβάλλον της Ευρώπης συνδέονται στενά με το πρόγραμμα Natura 2000 και το LIFE. Εάν λοιπόν θέλουμε να πετύχουμε τους στόχους μας στην στρατηγική βιοπικιλότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα είναι αναπόφευκτο να βρούμε πόρους για προγράμματα διατήρησης της φύσης όπως είναι το Natura και το Life. Όπως είπε ο Πρόεδρος, το πρόγραμμα LIFE αντιπροσωπεύει πολύ μικρό ε, μέρος του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιστεύω ότι κάθε σέντ που δαπανούμε για την ε, διατήρηση της φύσης ε, συμβάλλει στην βιωσιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της Επιτροπής για το σχέδιο γνωμοδότησής του. Θα ήθελα όμως να σταθώ σε κάποια σημεία που κατά τη γνώμη μου είναι σημαντικά. Καταρχήν, το θέμα των ε, χρηματοοικονομικών μηχανισμών. Αντιλαμβάνομαι την ανάγκη θέσπιση και εφαρμογή περιβαλλοντικών πολιτικών στην Ένωση και σίγουρα αυτοί οι μηχανισμοί ε, συνοδεύουν τα σχέδια. Αλλά προσοχή, γιατί ακόμη και το επενδυτικό σχέδιο του Juncker, το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, δεν είναι και πολύ ικανοποιητικό. Και αν ζητούμε μετάθεση σημαντικών κονδυλίων σε ένα κακοσχεδιασμένο ευρωπαϊκό πρόγραμμα από τα κράτη-μέλη, θα με βρείτε αντίθετη. Ε, θα πρέπει να επιτρέψουμε στις διοικήσεις και τα κράτη-μέλη, δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε ε, στα κράτη-μέλη, στις τοπικές αυτοδιοίκησεις ε, να διωγγώσουν τους προϋπολογισμούς τους ε, ή αν θέλουμε να ενισχύσουμε κάποιες ε, σιδηροδρομικές γραμμές ή γραμμές μετρό σε κάποιες πόλεις υπό το πρόσχημα του αγώνα κατά των κλιματικών αλλαγών και πάλι θα, θα σταθώ κατά της επικουρικότητας. Ε, και προσοχή, προσοχή με τις κλιματικές αλλαγές. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούμε τα δισεκατομμύρια ευρώ των φορολογουμένων των κρατών μελών για να χρηματοδοτήσουμε μια περιβαλλοντική πολιτική, περιβαλλοντική πολιτική για το κλίμα που μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υιοθετήσει και κανένα, καμία μια άλλη χώρα, παρόλο που παγκοσμίω υπάρχουν άλλε χώρε που ρηπαίνουν πολύ περισσότερο. Δεν μπορούμε έτσι ελαφρά την καρδία να κατασπαταλούμε χρήματα των φορολογουμένων. Και σε ό,τι αφορά του οργανισμού. Δεν μπορούμε να ε, με εμφόμαστε ε, τις περικοπές ε, σε οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους όταν το ίδιο πετούμε από τα κράτη-μέλη. Και οι οργανισμοί που αφορούν θέματα αρμοδιοτήτων μας συμφωνούν ότι θα πρέπει να μειωθούν στους πόρους τους περισσότερο από τους υπόλοιπους οργανισμούς. Η διαιτησία και η επιλογή θα πρέπει να είναι πιο σαφής και διαφανής. Γιατί αν θα θυσιάσουμε ένα τομέα εις βάρος του άλλου θα πρέπει να ξέρουμε γιατί το κάνουμε μετά από εμβριθή συζήτηση. Τέλος, όταν μιλούμε για κατάλληλους πόρους ε, θεωρώ ότι θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και σε καμία περίπτωση μια οικονομική αυτονομία ή μια άγουσα προς τους ε, ίδιους πόρους. Θα ήμουν κατά. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να σχολιάσει ιδιαίτερα το θέμα των οργανισμών, γιατί Κάποιοι είπαν ότι ε, στην πρόταση κάποιες ε, περικοπές που προτείνεται δεν ευθυγραμμίζονται με τις ε, δικές μας επιθυμίες και προτεραιότητες. Ναι, σε ό,τι αφορά τους οργανισμούς έχουμε πλήρη επίγνωση της δυσκολίας του έργου. Όχι μόνο των οργανισμών, αλλά και των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προς το παρόν πάντως, οι μειώσεις του προσωπικού καλύπτονται από μια διαδικασία streamlining ε, στους οργανισμούς. Δηλαδή γίνεται ανακατάταξη των υπαλλήλων προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι πραγματικές ανάγκες των οργανισμών. Και σε ό,τι αφορά τον προπολογισμό και το προσωπικό που προβλέπεται στους οργανισμούς, είναι θέματα που συζητήθηκαν ε, και στους ενδιαφερόμενους οργανισμούς και είμαστε πεπισμένοι ότι υπάρχουν πόροι που επιτρέπουν στους οργανισμούς να ανταπεξέλθουν στο έργο τους. Μετά τι ε, δραστηριότητε για τα βιοκτώνα της ε, ε, ΕΚΑ υπάρχει ένα πρόβλημα. Εκεί υπάρχει αλλαγή στο επίπεδο των τελών που θα λάβει η ΕΚΑ, ο αντίστοιχο οργανισμός και αυτό ίσως επηρεάσει τους μελλοντικούς πόρους και ίσως δημιουργήσει πρόβλημα στην διεξαγωγή του έργου. Αλλά θα πρέπει να μελετήσουμε τα στοιχεία για να δούμε ποιες είναι οι πραγματικές συνέπειες αυτής της αλλαγής. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω άλλον συνάδελφο να ζητά το λόγο. Να σας υπενθυμίσω το χρονοδιάγραμμα. 17 Ιουλίου τροπολογίες, διορία για τις τροπολογίες. 3 Σεπτεμβρίου θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή και στην Επιτροπή Προϋπολογισμών 3 ε, Σεπτεμβρίου λήγει η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Ενώ η ψηφοφορία στην Επιτροπή Προϋπολογισμών θα γίνει στη συνεδρίαση της 22ης-23ης Σεπτεμβρίου. Η ψηφοφορία στην Ολομέλεια θα γίνει κατά πάσα πιθανότητα στη δεύτερη Ολομέλεια του Οκτωβρίου. Αυτά μπορούμε να ολοκληρώσουμε τη συνεδρίαση και θα τα ξαναπούμε το απόγευμα. Γεια σας, καλώς μεσημέρι.